Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς την πρώτη τη επιτροπής ε, Φρανστήμενου στην επιτροπή μας που ήρθε στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Και μια που έχετε οριζόντες αρμοδιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα θέλαμε να μας πείτε μια, για τη γενική προσέγγιση σχετικά με την βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα πέστε μας τα σχέδιά σας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις ιστορικές πολιτικές και όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο έχει μια αντιπροσωπεία από την ΕΝΒΗ και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Και τον Ιούλιο θα παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ και εκεί θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί στη δουλειά μας για τους στόχους αυτούς και επειδή είναι πολύ προβεβλημένη αυτή η πρόταση, θέλουμε να ακούσουμε τι γίνεται με το πλαστικό μιας χρήσης και επίσης τι ισχύει όσον αφορά την κυκλική οικονομία και το σχετικό σχέδιο δράσης ή πρόγραμμα δράσης. Έχουμε επίσης το θέμα των εφαρμοστικών και κατεξοδοσίων πράξεων. Έχουμε προστείλει το Συμβούλιο μεταλλαγμένα, εκπομπές αυτοκινήτων και όλα αυτά είναι πραγματικά ένας φραγμός όσον αφορά το πώς θα προχωρήσουμε νομοθετικά. Ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε και έχετε το λόγο για ε, μας κάνετε μια εισήγηση και στη συνέχεια θα έχουμε συντονιστές και συναδέλφους που θα προβούν σε πρώτες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η εντολή σας αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, βιοποικιλία, βιοπικιλότητα ε, και θέλουμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε τη Συμφωνία των Παρισιών για το κλίμα. Πρόκειται για μεγαλύτερε προκλήσει τη εποχή μα. Να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ του ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τι συνθήκε διαβίωση και κανεί να μην μείνει απ' έξω. Για αυτή την μετάβαση στην βιωσιμότητα να εκμεταλλευτούμε τι συνεργείε ε, του θεματολίου 2004 και των Παρισίων. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει να κάνει με αυτούς τους στόχους μας που αλλιώ, αν δεν κάνουμε όλα αυτά που είμαστε, δεν μπορούμε να του πετύχουμε. Και είχαμε το έγγραφο προβληματισμού, το οποίο δημοσιοποιήσαμε για τη βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030. Και με χαρά μου διαπιστώνω ότι οι προτάσει μα για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο αναβαθμίζουν τι πολιτικέ για το κλίμα και αυτό διαπνέει όλο τον προπολογισμό. Επίση, είπαμε ότι θέλουμε τη θέσπιση κάποιων ε, εργαλείων που θα διέπουν ε, το Ταμείο Συνοχής και όχι μόνο για να κινητοποιήσουμε κεφάλαια σε βιώσιμες επενδύσεις. Γι' αυτό έχουμε μια σειρά νομοθετημάτων για βιώσιμη χρηματοδότηση και αυτά τον περασμένο μήνα. Το πρόγραμμα δράσης του Δεκεμβρίου του 2015 για την κυκλική οικονομία είναι success story, είναι ένα παράδειγμα προς τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Πάνω από 85% των μέτρων έχουν πιάσει τόπο και η πετυχημένη συνεργασία με τα θεσμικό και ιδίω την Επιτροπή σα, το Κοινοβούλιο γενικότερα έκαναν την διαφορά και έτσι προωθήσαμε τη σωστή νομοθεσία, όπω α πούμε για τα απόβλητα τον Απρίλιο. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και για τις ε, υπόλοιπε προτάσεις όπως για τα πλαστικά, προτάσεις επιτροπής, πολύ σημαντικά για τον κόσμο και επίσης για το νερό, το live και στα κράτη-μέλη αυξάνεται το ενδιαφέρον και στον ιδιωτικό τομέα και στου πολίτε για την κυκλική οικονομία και είναι πρωταγωνιστής η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την ε, μετάβαση. Και εδώ και παγκόσμια. Ε, ένα καινούριο πρότυπο για το περιβάλλον, για την οικονομία, και για την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον. Στρατηγική για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία είναι ένα όραμα. Έτσι, η βιομηχανία πλαστικών θα γίνει η ευφιέστερη, η πιο καινοτόμα, η πιο βιώσιμη παγκοσμίω. Μόνο 6% χρησιμοποιείται πλαστικό σε νέα προϊόντα με τη στρατηγική, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση πρόκειται να αποτελέσουν τμήμα τη λυσίδα παραγωγή και θα είναι προσθεμένη αξία αυτό και θα βρει και απασχόληση. Γιατί λένε για περισσότερο πλαστικό υπάρχει στον ωκεανό και είναι μεγάλο το κόστο, άρα χρειάζεται να υπάρξει ένα νομοθέτημα και αυτό είναι επιτακτικό, να έχουμε κάποιου κανόνε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα μέτρα, αυτά τα οποία αφορούν τα πλαστικά, όσον αφορά επίσης ε, αλληλευτικά εργαλεία εγκαταλειμμένα, οπότε έτσι ε, έχουμε 70% του συνόλου των απορριμμάτων στη θάλασσα, άλλα μέτρα, το καθένα για κάθε προϊόν και θέλουμε όλα αυτά να είναι σε προσθέστη τιμές στην αγορά. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει αυτή ε, μετάβαση, θα πρέπει αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο εύκολο. Αυτό και πασχίζουμε πρότασή μας. Είναι κορυφαία προτεραιότητα το τι θα γίνει με τα πλαστικά στις ε, παραλίες, τα καλαμάκια, πλαστικά πιάτα. Όλα αυτά ε, επιδέχονται εναλλακτικέ λύσεις από πιο βιώσιμα υλικά. Για κάποια αντικείμενα χρειάζεται και θεσία για αλλού χρειάζονται μέτρα, να υπάρχει συνδυτοποίηση, εθελοντισμός και επίσης ε, να είναι ευξημένη η ευθύνη του παραγωγού και να καλυφθεί το κόστος του καθαρισμού που τώρα το φέρει το δημόσιο, δηλαδή ο φορολογούμενος. Επίσης, χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει με τα μπουκάλια, τι θα γίνει με τα καπάκια, τα, ε, εκεί που βάζουν το φαγητό τέλο πάντων, τους περιέκτες ε, τροφίμων, τα υλικά ψαρέματος, οπότε θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα μέτρα και οπότε τα πλαστικά έχουν κόστος που το διαχειριστούμε και αυτό θα πλαισιωθεί από τους παραγωγούς και του πλαστικού και των εργαλείων αλίας. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι είναι κατεπήγον. Πριν το τέλος της εντολής να εγκριθεί αυτή η πρόταση πρέπει να βιαστούμε. Υπάρχει υποστήριξη του κόσμου για όλα αυτά. Θα ήταν ντροπή εάν δεν καταφέρναμε μαζί και τον Μάιο είχαμε καλές ε, ειδήσει και τον επόμενο Μάιο επίσης θα είναι ένα ορόσημο πριν τις εκλογές. Θα ήταν πολύ καλό. Διαρκούν ακόμα για τον κανονισμό των λοιπασμάτων οι διαπραγματεύσει. Πρόγραμμα δράσης και εκεί και Και οικονομία και θα πρέπει να ανακτώνται τα πλαστικά υλικά ε, αυτά που έχουν σχέση με τα λοιπάσματα πρότυπα αυστηρά ούτως ώστε να υπάρχει βιοδιαλυτότης και να προστατεύεται το νερό σε κάθε μορφή του. Είναι λοιπόν βιοδιασπόμενα αυτά τα πλαστικά εγκατακλείδη. Είναι ξεκάθαρο ότι το μακρόπνο κόστος καταστροφής του περιβάλλοντος είναι πολύ πιο μεγάλο από το βραχυπόδοσμο κόστος κάποιου φιλόδοξου κανονισμού. Εφτά από τους 10 βασικούς κινδύνους έμεσα ή άμεσα σχετίζονται με το περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορεί να λυθούν μόνο με την περιβαλλοντική πολιτική. Αν κάποιο μιλά για μόλυνση τη ατμόσφαιρα, πρέπει να μιλά και για κινητικότητα. Και για βιοποικιλότητα πρέπει να μιλά και για γεωργία και για πλαστικά των ωκεανών. Θα πρέπει κανεί να τα συζητά λαμβάνοντα υπόψη πώ καταναλώνουμε και πώ παράγουμε. Οπότε έτσι έχουμε νέους τρόπους συνεργασίας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα success story στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας στα πλαίσια ε, τη πετυχημένη χρηματοδότηση. Θα συνεχιστεί η προσπάθειά μα και στην επόμενη θητεία, με χαρά μου χρειαστώ μέσα και τότε, στην επόμενη θητεία και τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Και ε, στην αρχή τη θητεία μα υπήρχε φόβο το αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε με τα πρότυπα, την απορρίθμιση για το περιβάλλον και για, τα, για, τη γενική πολιτική και τελικά αποδείξαμε σε όλους όσους φοβόντουσαν ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται. Γιατί προοδεύσαμε σημαντικά και αποδείξαμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την οικονομία σου, γιατί μπορεί να είναι πρωτομιστρία η Ευρώπη. Σήμερα συνάντησα Καναδούς, εκπροσώπους από τον ΟΗΕ και αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος που υπόσχεται πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Βαλεάν. τρόποι συνεργασίας όπως είπατε. Ε, αυτό πασχίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και με τις άλλες επιτροπές, γιατί χρειάζεται να συνεργαστούμε παραπάνω. Βέβαια τα θέματα όλα αυτά είναι ελέγχτα για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μεγάλα πράγματα για τα, τα μικρά πράγματα και για τα πλαστικά. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να έχουμε ένα καλό Αποτέλεσμα, έχω τον παραδοσιακό κατάλογο των συντονιστών ή των εκπροσώπων τους που θα πάρουν το λόγο. Να ξεκινήσω με τον κύριο Λίζα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου που τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή μας και σε εσά. Στην αρχή είχαμε κάποιες αναταράξεις, αλλά τελικά το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ερώτηση όσον αφορά ε, τον τρόπο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε λάβει πάρα πολλές προτάσεις της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το αίτημα να ε, τα διεκπαιρεώσουμε πριν τι ε, ευρωεκλογέ. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένη ε, και τη διαθεσιμότητας των διερμηνέων για τους τριμερεί διαλόγους. Θα σας παρακαλούσα στις υπηρεσίες της Επιτροπής να πείτε ότι δεν μπορείτε να ασκήσετε τόση πίεση στο Κοινοβούλιο. Ε, κάπου υπόθηκε ότι δεν χρειάζεται ε, να διαβουλευτούμε με τους ε, ενδιαφερομένους, τους stakeholders. Αλλά θα πρέπει να έχουμε διαβουλεύσεις με τους ανθρώπους που θέλουμε να ακούσουμε προτού προχωρήσουμε στις εργασίες μας. Το άλλο θέμα είναι ότι στην, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια ιδέα που δεν ε, έχει ε, εγκριθεί επίσημα, ε, να μην υποβληθούν άλλες προτάσεις, το οποίο όμως σημαίνει ότι επί δύο χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμα και για θέματα σημαντικά, διότι μέχρι το τέλος της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα λάβουμε νέες προτάσεις και δεύτερον η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμεινο για να αξιολογήσει τα θέματα και να διαμορφώσει τις δικές της θέσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία ήδη επίγουν, ένα που με ενδιαφέρει ε, ιδιαίτερα είναι η ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ε, για τους ανθρώπους. Ε, νομίζω ότι αυτό επίγει. Σας παρακαλώ, ξεκινήστε λοιπόν με την μελέτη αντικτύπου και υποβάλλετε μας πρόταση όσο γίνεται πιο γρήγορα, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παλούτσιο από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε ικανοποιημένοι που η Κομισιόν, υιοθετώντα και τις δικές μας, τα δικά μας αιτήματα, παρουσιάζει διάφορες νομοθετικές προτάσεις. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο να είχαμε μια πιο τακτική εργασία που θα είχε αποφύγει αυτή την ε, υπερβολική παραγωγή νομοθετημάτων στο τέλος της θητείας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε και τα κείμενα. Τώρα, σε σχέση με την οδηγία για τα πλαστικά μονής χρήσης, ε, θα κάνουμε την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση εντός της θητείας. Θέλουμε ε, και το Συμβούλιο ε, ουσιαστικά να δράσει για τα πλαστικά. Μόνο στις χρήσει, θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις. Ε, το σενάριο που ορίζεται από την Κομισιόν ε, μας ε, οδηγεί στο να θέσουμε ένα καταστός για 10 χρόνια. Ε, χρειάζεται χρόνο. φτάνει αυτός ο χρόνος για να γίνει περαιτέρω έρευνα και να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις. Δεν πιστεύεστε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Δεύτερον, για κάποια είδη προϊόντων, ε, στο α του παραρτήματος ε, προβλέπεται από την οδηγία σημαντικές μειώσεις ε, και τα κράτη θα ορίσουν τους στόχους ε, για να υπολογίσουν τις διάφορες μορφές. Χρειάζονται στοιχεία για τα σημεία αφετηρίας και στη συνέχεια συγκεκριμένες μεθοδολογίες για την επίτευξη του στόχου. Δεν πιστεύετε ότι στο θέμα αυτό το κείμενο θα πρέπει να βελτιωθεί Επίσης, σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνεται από την Κομισιόν δεν φαίνονται αρκετοί. ιδίως η αναφορά στο στόχο της αποσύνδεσης της ε, ε, οικονομικής ανάπτυξης με την ε, κατανάλωση των πρώτων υλών, όπως και με το θέμα των πράσινων κρατικών προμηθεών. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τη γνώμη σας και για αυτά τα θέματα, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βυσνιεύσκα από το Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Η έκθεση για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφόρα ανάπτυξη που θετήθηκε τον ε, Ιούλιο λέει ότι η επίτευξη των στόχων εξαρτάται από τρεις πυλώνε. Χρειαζόμαστε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς ε, παράγοντες. Αυτοί οι τρεις πυλώνε είναι πολύ σημαντικοί. Επίσης, όταν συζητήσαμε την οδηγία ETS για την εμπορία εκπομπών, είπαμε ότι μια κλιματική πολιτική έχει Οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, αλλαγές ε, στα πλαίσια ε, της COP24. Περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν για τη μικροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα. Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την αλληλοεξάρτηση μεταξύ του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού πυλώνα. Και η δεύτερη ερώτηση τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες ε, που εξαρτώνται πολύ από τα ορυκτά καύσιμα, ε, παραδείγματο χάρη στον Άνθρακα, Εσλεσία και άλλες περιοχές μπορούν να τύχουν τις υποστήριξεις της Κομισιόν και τις κατανόησης της Κομισιόν ε, στα πλαίσια αυτής της νέας μακροπρόθεσμας κλιματικής στρατηγικής. Άλλη ερώτηση, μείωση του διοξιδίου του Άνθρακα στις μεταφορές. Εδώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ παρουσιάζει τις προτάσεις της για τις μειώσεις διοξιδίου του άνθρακα στις μεταφορές, ε, γιατί δεν παρουσιάσετε μια λεπτομερή ανάλυση, μια λεπτομερή μελέτη αντικτύπου και ποιο είναι ο αντίκτυπο ε, της πρότασης αυτού ε, στα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλότερο κατακεφαλία ΑΕΠ. Άλλη ερώτηση. Έχετε κάποια σχέδια για το πώς ε, θα υποστηρίξετε τις πιο στοχές χώρες ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση ή απλώς ε, παθητικά θα περιμένετε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Άλτε, η κυρία Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, δεν σκεφτόμουν να πάρω το λόγο σε συντονίστρια και καθώς ε, είναι διαθέσιμο το σλότ, ε, ζήτησα το λόγο. Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά απευθυνόμαστε στην Κομισιόν. Είχαμε αναφερθεί και στο θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών εδώ βρισκόμαστε στο τέλος, πριν το τέλος ε, να πρέπει να τρέξουμε μέσα στο χρόνο και να λύσουμε αρκετά πολύπλοκα πράγματα. Θα το κάνουμε βέβαια και ιδίω ε, για το θέμα των πλαστικών ε, ε μιας χρήσης. εδώ ε, συναντούμε διάφορους, αλλά όλοι αναφέρουν την ίδια ανησυχία, ότι είναι πολύ ο χρόνος. Ήθελα να το υπογραμμίσω κι εγώ και ίσως να ακούσουμε και τον κύριο Τίμερμανς ε, θα έχουμε στα τέλη Αυγούστου να μπούμε στην καρδιά της οδηγίας και στο κείμενο που μας προτείνεται, όμως θα θέλαμε να σας ακούσουμε σε σχέση με την παγκόσμια διάσταση. Γνωρίζουμε όλοι τα αριθμητικά στοιχεία, είναι τρομακτικά ε, και η ζημία που προκαλείται από τα πλαστικά, ε, κυρίως στα θαλάσσια οικοσυστήματα, κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ετησίως. Ακόμη και αν είχαμε 100% ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ δεν θα άλλαζαν τα πράγματα. Ποιο είναι το περιθώριο στο παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ε, ξέρουμε ε, ότι τα κύρια προβλήματα υπάρχουν ε, στην Ασία ποιος είναι ο τρόπος που θα, αρθρώσουμε αυτή τη διπλωματία των πλαστικών, τι θα κάνουμε στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι τα δικά μας όπλα και τα εργαλεία για να το πράξουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όκεν από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Τίμερμανς. Ιδιαίτερα που αναβάθμισε το θέμα των πλαστικών. Από τα μικρά πράγματα στα μεγάλα πέρασε το θέμα αυτό. Ε, αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου και όπως είπατε και εσείς ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ε, ξεκινήσουμε επικοδομητική συζήτηση σχετικά με ε, τα ε, πλαστικά μιας χρήσης, αλλά η όλη συζήτηση ε, σήμαινε ότι δεν ε, μπορέσαμε να έχουμε ολοκληρωμένη απαγόρευση των ε, οξυδιασπόμενων, διότι είναι πολύ επιθετική η εκστρατεία υπέρ των πλαστικών αυτών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ε, χρειάζεται λοιπόν πολύ ισχυρή απαγόρευση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όσον αφορά τα κανονικά βιοδιασπόμενα, διότι αν βρίσκονται παντού στη φύση και απαιτούν χρόνο για τη διάσπασή τους, αυτό είναι κακό. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε απλά αντικατάσταση των παλαιών ε, πλαστικών με τα βιοδιασπόμενα. Ε, θα ήθελα όμως και ένα πολύ σαφές μήνυμα όσον αφορά τα οξοβιοδιασπόμενα. Ε, ο πρόεδρος Ιούνκερ είπε ότι θα δημιουργήσει ειδική ομάδα Task Force που θα εξετάσει το θέμα της επικορικότητας. Ακούσαμε ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ έχει μία πρόταση επανεθνικοποίησης της έγκρισης ε, των ζυζανιοκτώνων και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αν συμβεί αυτό, αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε νομοθεσία. Ήδη είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμίσει κανείς ε, τα φυτοφάρμακα. Είχαμε κάποια πολύ βαριά θέματα για τα έντομα, για τις μέλισσες, ε, λόγω ακριβώς των ε, φυτοφαρμάκων. Εάν λοιπόν ε, το θέμα αυτό επιστρέψει σε εθνικό επίπεδο, δεν θα έχουμε πια νομοθεσία και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό θα είναι εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητας. Σας παρακαλώ λοιπόν υποσχεθείτε μου ότι δεν θα δεχτείτε κάτι τέτοιο. Υποσχεθείτε μου ότι αυτό θα παραμείνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να έχουμε μέλλον χωρίς επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μερικές φορές οι ερωτήσει είναι πιο τεχνικής φύση. θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θα ήθελα όμως να ε, τις ε, μεταφέρω και στους συναδέρφους μου ε, που είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Να ξεκινήσω όμως ε, από το θέμα της επίγουσας δράσης. Σίγουρα δεν αποτελεί πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πιέσουμε αδικαιολόγητα τους ευρωβουλευτές. Πιστεύω όμως ότι λίγος χρόνος απομένει και Έχουμε μεγάλο όγκο ε, νομοθετικών σχεδίων ε, στα γραφεία μας ε, και έχουμε επίσης μεγάλο όγκο δουλειάς στο Συμβούλιο. Στις ευρωεκλογές του χρόνου καλό θα είναι να παρουσιάσουμε αυτά που έχουμε κάνει. Αυτό θα εντυπωσιάσει πολύ περισσότερο στους ψηφοφόρους μας από τις υπέροχες προτάσεις μας. Στα μάτια των ψηφοφόρων μας, Είμαστε ένα σώμα, δεν θα κάνω τη διάκριση. Δεν θα πούνε ότι α, το Κοινοβούλιο έκανε καλή δουλειά, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε καλή δουλειά και όχι ε, το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρώπη ενεργεί και εμεί ε, αποτελούμε μέρο τη Ευρώπη. Γι' αυτό και εγώ και οι συναδελφοί μου ε, νιώθουν ε, ότι κάποια θέματα επήγουν και πρέπει να ολοκληρωθούν ε, μέχρι το τέλο τη θητεία μα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υποβάλουμε άλλε προτάσει. Όχι, σημαίνει όμω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θέματα που δεν έχουν προταθεί μέχρι σήμερα, μάλλον δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της θητείας. Εάν λοιπόν υποβάλλουμε προτάσεις τώρα, ουσιαστικά υποβάλλουμε προτάσεις προς το νέο κοινοβούλιο, το επόμενο κοινοβούλιο ή την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτή λοιπόν την αίσθηση του κατεπήγοντο, ε, δεν λέω ότι δεν θα υποβάλουμε νέε προτάσει, αλλά καλώ του συναδέλφου μου στο Σώμα των Επιτρόπων να δεσμευτούν προσωπικά, να συμμετάσχουν στους τριμερεί διαλόγους, στις συζητήσεις, ώστε να φροντίσουμε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μην ε, κατηγορηθούμε ότι δεν κάναμε αρκετά για να ολοκληρώσουμε κάποια θέματα. Φυσικά είναι ελεύθεροι οι ευρωβουλευτέ όσον αφορά την ε, εντολή τους. Το ίδιο ισχύει για το Συμβούλιο. Τελικά όμως όλοι μας θα κριθούμε, θα επενεθούμε ή θα κατηγορηθούμε για τα αποτελέσματα που θα έχουμε πετύχει ή δεν θα έχουμε πετύχει. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά. Μιλάμε για το θέμα της μικροβιακής αντοχής, υποθέτω. Ε, πέρσι υιοθετήσαμε το σχέδιο δράσης για την ενιαία υγεία. Στρατηγική προσέγγιση για τα φάρμακα είναι μία από τις δράσεις που έχουν ε, αναφερθεί στο πλαίσιο αυτό. Είναι λογικό να συνδέσουμε μεταξύ τους τα δύο αυτά θέματα. Ε, αντιβιωτικά ε, έχουν βρεθεί στο νερό και στη, στο έδαφος ε, και γι' αυτό η πιο φρόνιμη χρήση των αντιβιωτικών ε, και η πιο φρόνιμη χρήση των ε, υγρών αποβλήτων ε, θα ήταν κάτι λογικό. Νομίζω ότι σήμερα ψηφίζεται πάνω στην έκθεση αυτή, έτσι δεν είναι. Ε, έχουν ε, υποβληθεί τροπολογίες στην έκθεση αυτή που έχουν να κάνουν με την στρατηγική προσέγγιση ε, εκφράζοντας κιόλα σε δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση. Και φαντάζομαι ότι το Σεπτέμβριο θα πάει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Εργαζόμαστε λοιπόν πάνω στην στρατηγική προσέγγιση για τα φάρμακα. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι είναι πολύ πλοκό το θέμα και πολύ τεχνικό και θα πρέπει να διαβουλευτούμε με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων για να φροντίσουμε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους δείκτες, πρόθεσή μου είναι διότι είμαστε σε επιφυλακή στο θέμα αυτό. Θα αλλάζουμε τους δείκτες όταν έχουμε νέα δεδομένα. Τους προσαρμόζουμε και τους επικαιροποιούμε συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, μείωση των ε, προϊόντων μιας χρήσης ε, και σχετική στόχη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε σχετική μεθοδολογία. Εάν όμως δεν κάνω λάθος, αυτό που έχουμε υποβάλει αυτή τη στιγμή είναι από ό,τι γνωρίζουμε με βάση όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα η καλύτερη λύση. Εάν όμως είναι σωστή η αίσθησή μου, η επιστήμη και οι αγορές κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει πάνω στα θέματα αυτά. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στις εξελίξεις. Γι' αυτό πιέζουμε τις αγορές, πιέζουμε τους επιστήμονες. Ε, θεωρούσαμε ότι τους πιέζουμε ε, όσο γίνεται, αλλά τελικά βλέπω ότι τα πράγματα εξελίσσονται ακόμα πιο γρήγορα. Εάν λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον και χρηματοδότηση, θα πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς. Όσο όμως είναι σωστή και διαμφισβήτητη η μεθοδολογία μα. νομίζω ότι η προσαρμογή σε νέες εξελίξεις είναι πιο εύκολη. Μπορούμε λοιπόν, κύριε Παουλούτσι, να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας εάν είναι απαραίτητο. Βλέπω να υπάρχει σχέση ανάμεσα σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές εξελίξεις. Σίγουρα αυτά συνδέονται μεταξύ τους άρρηκτα για να βελτιώσουμε το περιβάλλον, στο παρελθόν θεωρείται κάτι ωραίο, κάτι καλό. Σήμερα είναι απαραίτητο. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μεγάλο λάθος εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στη βιωσιμότητα και τα κοινωνικά θέματα ή τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για τη βιωσιμότητα δεν μιλάμε μόνο για το περιβάλλον, Μιλάμε και για την κοινωνική βιωσιμότητα. Ε, πού θα βρίσκονται οι θέσεις απασχόλησης στο μέλλον δεδομένης ε, της ε, ρομποτοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε αρκετά ευφυείς και ευπροσάρμοστοι ώστε να φροντίσουμε στο μέλλον ο κόσμος να έχει δουλειές πώς ε, θα διασφαλίσουμε την ενεργειακή μετάβαση και τη μετάβαση στους τρόπους μεταφοράς, ε, πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Αυτά είναι απαραίτητα για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να πω το εξή και να είμαι απόλυτα σαφής. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Εάν δεν προσαρμοστούμε, ε, θα αναγκαστικά θα θα υποφέρουμε, θα δεχτούμε πολύ αρνητικές ε, συνέπειες λόγω της ε, αλλαγής του κλίματος. Τα πλαστικά αποτελούν το τέλειο παράδειγμα της κατάστασης αυτής σήμερα. Δεν γνωρίζουμε καν ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην υγεία μας και τα μικροπλαστικά υπάρχουν παντού ε, στα πιο βαθιά σημεία των ωκεανών μας, στα σώματά μας, στο μπουκάλι αυτό που κρατάω. Το 90% του εμφιαλωμένου νερού περιέχει μικροπλαστικά. Και δεν μιλάμε για κάτι που είναι πολυτέλεια, κάτι που θα ήταν ωραίο να κάνουμε. Μιλάμε για πράγματα που είναι απαραίτητο να γίνουν. Ε, και θα επανέλθω στα πλαστικά τύπου όξο σε λίγο. Ε, είναι θέματα που θα έχουν τεράστιες συνέπειες στο μέλλον μας. Ε, και ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να εξελιχθούμε ε, να έχουμε πιο βιώσιμο μέλλον ε, και νομίζω ότι είμαστε το μέρος του κόσμου που θα καταφέρει να κάνει τη μετάβαση αυτή πιο γρήγορα όσον αφορά την ροποτοποίηση και την ψηφιοποίηση και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει αυτή την πεποίθησή μας να πείσουμε τους ανθρώπους της Ευρώπης ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έχουν θέση σε αυτόν τον ε, νέο κόσμο. Πιστεύουν ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να υπερασπιστούν ε, την, ε, τις ε, συμβατικέ λύσει. Θα είναι όμως τραγικό και ιστορικό σφάλμα εάν εμεί ω πολιτικοί δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους μας ότι η μετάβαση αυτή θα γίνει και καλύτερα να ε, συμμετέχουμε και εμείς στη μετάβαση αυτή. Όσον αφορά τις μελέτες αντικτύπου, ε, Ήδη απάντησα στο θέμα της έλλειψης χρόνου. Επίσης, όσον αφορά τα πλαστικά, είχα σήμερα το πρωί συνάντηση με προσώπους ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, της Κίνας ε, και του Καναδά. Με μια στρατηγική για τα πλαστικά και ιδιαίτερα καθαρίζοντας τους ωκεανούς μας, έχουμε ε, συλλάβει το πνεύμα όλου του κόσμου. Αυτό είναι τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ασία. Και πολύ σωστά υπόθηκε ότι η συμβολή της Ευρώπης στο θέμα αυτό είναι σχετικά μικρή. Εάν ε, όμως η Ευρώπη συμβάλλει στη λύση, θα είναι τεράστια η συμβολή μας, διότι και οι Κινέζοι αναζητούν λύση και γνωρίζουν ε, ότι επηρεάζεται η αλληλεία τους, ο τουρισμός τους, η υγεία τους, επειδή δεν υπάρχουν λύσεις στα θέματα αυτά. Ακόμα λοιπόν ε, και εάν η συμβολή μας στο πρόβλημα είναι σχετικά μικρή, παρότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στη δική μας υγεία και στο δικό μας φυσικό περιβάλλον, κοιτάξτε τις ακτές μας, βούτυξτε στις ευρωπαϊκές θάλασσες ε, και δείτε τι θα βρείτε κάτω ε, από την επιφάνεια της θάλασσας εγώ. Ε, από προσωπική μου πείρα μπορώ να σας πω ότι είναι συγκλονιστικά αυτά που βλέπει κανείς μπορεί σε απόλυτε τιμέ να είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη όμω βρει το κλειδί για βιώσιμε λύσει, τότε ε, ο αντίκτυπο των λύσεων αυτών ε, θα είναι τεράστιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και για την Ασία. Και βλέπουμε πώ αντιδρά η Ασία στα σχέδια μα Και μάλιστα όχι μόνο οι πιο αναπτυγμένε χώρε. Είδα ενθουσιώδει αντιδράσει από την Ινδονησία, από την Κίνα, που ανέφερα ήδη, από την Ταϊλάνδη από όλε τι χώρες αυτές που βλέπουν ε, ότι ε, ο τουρισμός και η αλεία τους, ε, οι σημαντικότεροι οικονομικοί τομεί τους επηρεάζονται και γι' αυτό αναζητούν λύση. Καλύτερη νομοθεσία, απαγόρευση των οξοπλαστικών. Όπως ανέφερα στην στρατηγική για τα πλαστικά και στο πλαίσιο του REACH, ε, προσπαθούμε να βρούμε ε, λύση και συζητάμε το θέμα της απαγόρευσης των οξοπλαστικών. Είναι λοιπόν θέμα που βρίσκεται στο θεματολόγιο μας και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία στο πλαίσιο του REACH. Θα σας ενημερώσουμε ε, σχετικά με τα αποτελέσματα όταν καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Η ειδική ομάδα Task Force για την επικουρικότητα. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα που ανεφέρατε. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου. Θα το εξετάσω όμως. Άλλωστε είμαι πρόεδρος ε, της ειδικής ομάδας αυτής, ε, άρα αποτελεί αρμοδιότητά μου. Θα το εξετάσω. Αυτά έχω να πω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. This... Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι φαίνεται αυτό το θέμα είναι πιο εύκολο από το θέμα του κλίματος, το να πείσουμε δηλαδή τις άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν. Η πιο εύκολη λύση είναι απλή απαγόρευση, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο. Για ένα λεπτό θα είναι ο χρόνος ομιλίας. Όποιος θέλει να μιλήσει, έχω κάποια ονόματα εδώ. Αλλά αν θέλετε κι άλλοι να ζητήσετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Γκρουστέτ, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον ε, πρώτο αντιπρόεδρο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι είναι κρίμα. Χάσαμε το πρώτο μισό αυτή τη θητεία. Είχαμε έναν επιβραδυμένο ρυθμό. Και σήμερα καταραίουμε από τη δουλειά, είναι κάπως αργά. Εμένα με εκπλήσει, δεν υπάρχει ε, ουσιαστικά κανένας χώρος σε σας για το θέμα της πολιτικής της υγείας, ε, όμως βλέπουμε ε, τις ε, συνέπειες, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τις πάνες θέσεις, την καταπολέμηση του καρκίνου, αυτό της αφορά όλους, η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, οι συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού και φυσικά το μέλλον της βιοτεχνολογίας. Όλα αυτά, αν δεν ε, μιλήσουμε για αυτά, είναι πολύ κακό το μήνυμα, είναι η παναχώρηση. Μιλήσατε για συγκεκριμένες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν απέναντι στο εκλογικό μας σώμα. Η πολιτική της υγείας για σας δεν υπάρχει. Και αυτό που με ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ότι τρέχουν διάφορες φήμες ότι την επόμενη φορά δεν θα υπάρχει αρμοδίος επιτρόπος για την υγεία. Πιστεύω λοιπόν ότι στη δική μας Επιτροπή Δημόσια Υγεία Περιβάλλον είμαστε πολύ άριθμοι όλοι εμείς που ζητούμε οπωσδήποτε η πολιτική της υγείας που είναι ουσιαστική πολιτική, ουσιαστική και για την ε, οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ισότητα όλων ε, απέναντι σε μια υγεία ασφαλή και προσβάσιμη από όλους χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει μια πολιτική εμφανής που δεν πρέπει να εξαφανιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δύο συγκεκριμένε σύντομε ερωτήσει. Για αυτή τη κεφαλιά που θα πρέπει να λύσουμε για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα, πρέπει για μη τοξικό περιβάλλον μέχρι το 2018 να έχετε μια στρατηγική. Όμως, δεν έχουμε υπόψη μας κάποιο είδους στρατηγική που προσεχώς θα εξαγγείλεται. Πέστε μας επομένως τι μέτρα θα πρέπει να λάβετε. Ο μιλητής μιλά πολύ μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούγεται καλά. Επίση τι γίνεται με τη στατική για τους ανδρογενικού διαταράκτε. Λέμε ότι έχει προετοιμαστεί και θα είναι τα τέλη του έτους έτοιμη. Και γι' αυτό θα να σας ρωτήσω τι γίνεται, πώς έχει η κατάσταση. Τι γίνεται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, σας ευχαριστώ. Thank you very much. Now... Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος Αλαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επιστρέψουμε στο θέμα της ε, στατικής για τα πλαστικά, γιατί το World Economic λέει ότι το 80% των πλαστικών στην θάλασσα ε, προέρχεται από 10 πηγές ε, βιδάτινε, 8 στην Ασία και 2 στην Αφρική, οπότε τελικά είναι πρωτοπόρα η, η Ευρώπη στη στρατηγική της καταπολέμησης ε, της χρήσης του πλαστικού. Αντικειμενικά όμως, ε, από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε κάνει και πολλά πράγματα για το τελικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε έχουμε σωστή προσέγγιση Άρα μήπω κάτι έχουμε ξεχάσει, γιατί υπάρχουν κάποιε τεχνικέ εναλλακτικέ, υπάρχουν εναλλακτικά υλικά και αυτά βέβαια μπορούν να συγκρατήσουν σε επιπτώσει το περιβάλλον. Ε, όχι χαρτί, αλλά κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε, κάτι άλλο μπορούμε να πετύχουμε. Και ας πούμε να τα σκεφτούμε σφαιρικά δεν λέω ότι πρέπει να σκοτώσουμε έναν παραγωγικό κλάδο ε, και από την άλλη μεριά να μην καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα για το περιβάλλον, για μια οικονομία που είναι συνδεδεμένη με το πλαστικό. Ευχαριστούμε. Κύριε Μελιόρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε και για τις παρατηρήσεις σας και θα επανέλθω στην ε, στρατηγική για τα πλαστικά μιας χρήσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό βήμα. Ανησυχώ όμως σχετικά με το πώς ε, θα μεταφέρει το μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καταφτάνει ως απαγόρευση στα κράτη-μέλη. Η ε, πολίτες ε, νιώθουν την απαγόρευση. Όταν το συζητάει κανείς όλοι λένε ναι, θα πρέπει να το έχουμε κάνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιώσιμα υλικά, αλλά η Ευρώπη ουσιαστικά απαγόρευση υιοθετεί. Και το πρωτόκολλο του Κιώτο σκοπό έχει να φέρουμε τους ανθρώπους με το μέρος μας και να τους υποστηρίξουμε. Επίσης, όσον αφορά την διπλωματία για την ε, πολιτική του κλίματος, ε, το ε, Κοινοβούλιο είχε μια κοινή συνεδρίαση και εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος συμμετείχαμε και σημαντικό είναι έτσι να μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σράγερ Πίρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, που βρίσκεστε εδώ. Καταρχάς, ε, η στρατηγική για τα πλαστικά είναι κάτι που υποστηρίζει πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε πει στον, στον ε, Υπουργό μας ε, τον Ιαν Μπρόγκα, ότι σα υποστηρίζουμε απόλυτα στο θέμα αυτό. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Αλία, συζητήσαμε το θέμα θα αποζημιώσουμε όλους τους αλληλείς που συγκεντρώνουν όλα τα απορρίμματα που βρίσκουν ε, στη θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα που ε, θίξαμε στην ε, Επιτροπή Αλίας. Πώς θα τους αποζημιώσουμε. Άλλο θέμα είναι η κυκλική οικονομία και η γεωργία. Πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για αυτούς τους τομείς. Η νομοθεσία από μόνη της ε, είναι δύσκολη. Γνωρίζετε τι γίνεται στις κάτω χώρες. Χρειαζόμαστε όμως ε, κάποιες κατευθύνσεις από την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κάποια μεταβατικά μέτρα που να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όμως όλα αυτά. Ε, και ο κύριος Κατάινεν ε, το έχει πει αυτό. Ε, υπάρχει όμως πολλή γραφειοκρατία που εμποδίζει τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαβία έχει δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Επιστρέφω, για ένα άλλο θέμα. Για τα κατάλοιπα των τροφίμων. Γιατί θέλουμε να βιώσουμε μια ανάπτυξη και βέβαια υπάρχει ως στόχος ε, το να μειώσουμε τη διασπάθηση αυτών των τροφίμων. Και είπαμε ότι με το 2030 πρέπει να τα έχουμε μειώσει αυτό το, το επίπεδο των απορριμμάτων στα πλαίσια αυτής της κυκλικής οικονομίας. Μπορείτε να μας πείτε σε σχέση με το πόσο κοντά είμαστε σε αυτούς τους στόχους, τι συνεργασία υπάρχει με τα κράτη-μέλη, με τους ΜΚΟ, τι γίνεται με την καμπάνια ευαισθητοποίησης, γιατί εύκολο είναι να θέτουμε στόχους με την νομοθεσία, αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή όλων. Αυτού του είδους η σπατάλη των ε, τροφίμων να μειωθεί. Θα πρέπει να γίνει αυτό προτεραιότητα στην Ένωση. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θέλει άλλο το λόγο. Όχι. Άνι, εκτός σειράς. Πρόεδρε. Το θέμα είναι αφού συζητήσαμε για την αλληλεία, να δούμε τι θα κάνουμε τη συμφωνία για το κλίμα. Τι γίνεται με τις μικρές οικογενειακέ εταιρείε. Ξέρετε πριν να πρόκειται και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια εύστοχη λύση για αυτόν τον κλάδο. So now it's up ο Επίτροπος. Για να αρχίσουμε από το τέλος, την τελευταία ερώτηση, να σας τα πω στα Ολλανδικά. Όσον αφορά την αλληλεία, δεν χρειάζεται να πείσετε εμάς να τα πείτε στους συναδέλφους σας, τους άλλους ευρωβουλευτές. για την αλία με ηλεκτρικό ρεύμα, ε, βεβαίω και έχει επιπτώσει στην υγεία μας. Είπαμε για τα μικροπλαστικά που καταναλώνουμε στα ρούχα, στο φαγητό, στο νερό, στην ατμόσφαιρα. Και μετά αυτά τα όξοπλαστικά, ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η επίπτωση στην υγεία. Δεν υπάρχει βιοπικιλότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για την υγεία μα και είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα που μα απασχολούν, στα οποία εμπλέκεται ο παράγον υγεία. Και η κυρία Γκροστέτ μα είπε ότι κάποιο ίσω από το ΕΛΚ είχε την ιδέα στην επόμενη επιτροπή να μην υπάρχει επιτροπή με χαρτοφυλακή υγεία. Τέλο πάντων, τώρα υπάρχει. Κανεί στην επιτροπή δεν σκέφτηκε, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Έχουμε για τα θέματα της, υγεία υγείας έναν ικανότατο συνάδελφό μου τον κύριο Τριοκάτης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα φτάσουμε στο σημείο. Αυτό. Μα το θέμα θα έχει αυξανόμενη και όχι μειωμένη σημασία. Από αλλού προέρχεται αυτή η ιδέα, όχι από εμά. Όσον αφορά τώρα την στατική, ναι, ξέρετε. Έχουμε εθνικές αρχές. Α, θυμάμαι στο Συμβούλιο. Ε, κάποια προεδρία έλεγε θα μειώσει τους επιτρόπους και δεν ξέρω αν θα υπάρχει επιτρόπος ε, υγείας στο μέλλον κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη τέτοιες ε, προτάσεις. Πάντως από εμά δεν προέρχονται. Σας διαβεβαιώ. Για τους ενδοκρινικού διαταράκτες πέρσι συγχωρούσαμε τα κράτη-μέλη για να δούμε με τι κριτήριο θα δουλέψουμε όσον αφορά την νομοθεσία για τα βιοκτώνα και τα ζυζανιοκτώνα και είπαμε ότι θα δουλέψουμε σε ένα σφαιρικό πλαίσιο για αυτούς τους διαταράκτες και εξετάζουμε τώρα πώς μπορούμε να επικαιροποιήσουμε την προσεγγίση μας, να λάβουμε υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις, τις διάφορες πλευρές, τις διάφορες πολιτικές, τη συνέπεια μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο. Ε, συνεχίζει την προσπάθειά μας. Και σας προτείνω, αν θέλετε, να τα πείτε με τον κύριο Αντριουκάκη, αφού τον καλέσατε. Πασχίζουμε και αφιερώνουμε πολλή ενέργεια σε αυτό το μέτωπο και ελπίζουμε να θα αποσπάσουμε κάποια αποτελέσματα. Το μη τοξική περιβαλλοντική στρατηγική. Πολύ περίπλοκη υπόθεση. Γίνονται διάφορε αξιολογήσει για τα χημικά. Οπότε δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια στρατηγική προ του τέλου τη θητείας. κοντά είναι το τέλος της διετίας οπότε δεν ξέρω αν αξίζει κανείς να βιαστεί. Πάντως, λαμβάνω υπόψη αυτό που είπατε. Βέβαια και θεωρείται σημαντική την υπόθεση αυτή. Βέβαια θα πρέπει να εξαγάγουμε από την ε, πρόσφατη εξολόγηση τα συμπεράσματα ε, για τα χημικά, για το fitness check και ακόμα θέλουμε να δούμε πώς θα ε, τα δημοσιοποιήσουμε όλα αυτά και οι εμπλεκόμενοι να έρθουν και να ξεκινήσουμε έναν διαρκή διάλογο για επίτευξη πρόοδου. Τώρα για απαγορεύσεις και τις οικονομικές επιπτώσεις. Να σας τα πω ομά. Τα περισσότερα δεν παράγονται καν στην Ευρώπη από αυτά τα προϊόντα, τα οξοπλαστικά. Να σας το πω έτσι, ως προσωπική εμπειρία, όσο αξίζει. Και αυτά 18 χρόνια ασχολούμαι ως πολιτικός με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, με τους πρώτους που τα χρησιμοποίησε και όταν είχαμε αυτά τα σχέδια με απαγορεύσεις και ε, πλαστικά μια χρήση Λέγανε πω από πάλι και άλλες απαγορεύσεις στις Βρυξέλλες. Τελευταία τετραετία. Η πιο δημοφιλής πρόταση που έγινε, η πιο δημοφιλής πρόταση ήταν αυτή ακόμα και από τα βρετανικά ταμπλόιντ. Γι' αυτό λέγαμε μπας και κάτι κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό σα λέω, η πρωτοβουλία για τα πλαστικά και η πρόταση για τα πλαστικά μια χρήση είναι από αυτές τι ιδέες που έρχονται και καμιά φορά είναι φανταστικές, αλλά καμιά φορά είναι πολύ πρόημε. Άλλοτε έρχονται στην ώρα τους. Ένα, ε, πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ε, στην ώρα της και πάρα πολύ πετυχημένη. Γιατί νομίζω πιάσαμε τον παλμό της κοινωνίας πάνω από το 80% των Ευρωπαίων δηλώνουν ε, ότι του αρέσει αυτό γιατί είναι για το περιβάλλον σημαντικό και όλα είναι και περισσότεροι. Καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει επιπτώσει θετικέ για την υγεία του. Μα λένε, τι, τι, λέτε, τι λέτε λέτε για τα καλαμάκια, λεπτομέρειε για τα, τα, αυτά που καθαρίζουμε τα αυτιά μα τι οδογλυφίδες, τις ειδικέ μα. Ναι, αλλά ε, είναι επιπτώσεις μεγάλες για την υγεία. Ακόμα και το McDonald's απαγόρευσε σε πολλές χώρες τα πλαστικά καλαμάκια. Δύο-τρία χρόνια υπήρχε μεγάλο ζεσταγμός. Τώρα το κάνουν. Άρα, άρα, να, σιγά σιγά ήρθε η αλλαγή. Οπότε δεν φοβάμαι ότι ε, οι απαγορεύσεις είναι φραγμός, είναι ε, φρένο. Όχι, όχι. Συνεχίζουμε και θα μας ευχαριστούν τώρα σαν τη διπλωματία την κλιματική πάρα πολύ σημαντική και προβληματίζουμε πάρα πολύ όσον αφορά το δυνές περιβάλλον. Αυτή τη, τη, νέα μορφή διπλωματίας που είναι κάτι σαν ένας νταΐς να συμπεριφέρεται και να λέει δεν με νοιάζει και λοιπά. Όχι, εγώ νομίζω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διπλωματία, θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την ρότα όπω ξεκίνησε στην Γαλλία προπαρασκευαστικά και να συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση σε Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Αυτή που είχαμε ε, μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι. Οπότε θα είμαστε πρωτοπόροι και θα μας ακολουθήσουν και άλλοι. Ακόμα κι αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν μας ακολουθήσει, πάρα πολύ στις ε, είπα πολιτείες, επιχειρήσεις, ε, δήμοι ε, μας ακολουθούν. Είμαι με αισιόδοξος. Α, για την Ελία τώρα. Θα έχουμε έξτρα δαπάνες το θέμα αυτό των αλληλευτικών εργαλείων. Όπου υπάρχουν πλαστικά, οι παραγωγοί φέρουν το βάρος του οικονομικό. Θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα φέρουν την ε, δαπάνη οι αλίες. Και το κόστος του κουραγός θα είναι 0,16% από τον ετήσιο τζίρο του κλάδου. Τώρα, οι ίδιοι πληρώνουν το κόστος της ε, μόλις στη θάλασσα. Γιατί ψαρεύουν πλαστικό με τα Ψάρια καταστρέφονται οι προπέλες των σκαφών. Ακριβώς λόγω του πλαστικού που κυκλοφορεί στη θάλασσα. Στα θαλασσινά, στα ψάρια, βλέπει ο κόσμος που πάει τα φάει πλαστικά και χάνει την εμπιστοσύνη του. Οπότε, όταν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη, χάνουν οι οικονομικά οι Κόστος 57 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα μειώσουμε το πλαστικό. Αυτό θα ωφελήσει όλο τον κλάδο. Οπότε την ευθύνη τώρα με την πρότασή μας θα την αναλάβουν οι παραγωγοί και θα επιβαρυνθούν λιγότερο οι αλληλείς. Πολύ σημαντικό. Επίσης, για το επόμενο ταμείο αλληλείας θα γίνει αυτό το οποίο είχε ζητηθεί. Θα υπάρχει επιδότηση στους ψαράδες που φέρνουν ε, υλικά πλαστικά στην ε, ξηρά. Κύριε Ραβία, σας ευχαριστώ για τη διασπάθηση των τροφίμων. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό που θίξατε. Εμείς αστιαζόμαστε στο πώς η τριτογενής νομοθεσία θα ολοκληρωθεί γέρος. Λέτε ότι πρέπει να εστιαστούμε προς τα εκεί. Να έχουμε κοινή μεθοδολογία για να αποτιμήσουμε πόσο είναι η διασπάθηση, ένα κοινό πλαίσιο για συγκρίσιμα δεδομένα στατιστικά. Αρχάς επομένου έτους, κατά το Μάρτιο, θα έχουν προχωρήσει. Όχι, δεν καθυστερούμε λόγω εκλογών. Μέχρι το Μάρτιο σας υπόσχομαι ότι αυτό το οποίο θέλετε θα υπάρχει. Α, και άλλη μια ερώτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Να, πώς να το πω. Αν δημιουργήσουμε αντίθεση μεταξύ περιβάλλοντος και εργασμένων στην Ήπεθρο, όλοι βγαίνουν χαμένοι. Θέλουμε βιώσιμο περιβάλλον, αλλά να υπάρχει συμμετοχή των Γιώργων. Ε, αυτοί είναι που θα σας εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα. Και αυτό ακριβώς προτάθηκε από τον Επίτροπο Γεωργίας. Αν μπορέσει η Επιτροπή σας να μας βοηθήσετε να γίνει όσο γίνεται πιο πράσινη η γεωργική πολιτική, ε, τότε θα έχετε ωφελήσει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπα στην αρχή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεσμευόμαστε απόλυτα να εργαστούμε για όλα τα θέματα που είναι επιπάτη, τάπητος και όλα όσα έλθουν ε, μέχρι τα τέλη της ε, θητείας μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Αντιπρόεδρε. Thank you very much. Bye-bye.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 So, dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε μαζί σας τις ε, κάρτες σας. Since I worked at, uh, until the Λοιπόν, ε, καθώς δούλευα μέχρι τις 4.30 ε, το πρωί στον ε, τριμερή διάλογο, σας δω συγγνώμη που έχω λίγο αργούς ρυθμούς σήμερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε διεκπαιριωτικοί. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, έχετε τις κάρτες για την ψηφοφορία. Βλέπω κάποιους που δεν έχουν, όπως η κυρία Γκαρντίνη. Μάλιστα, τώρα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ηλεκτρονικά η πρώτη ψηφοφορία αφορά τον συμβιβασμό για την ε, πρόταση που αφορά τη θέσπιση κοινωτικών διαδικασιών χορήγηση άδεια και υποπτία όσον αφορά τα φάρμακα προ για ανθρώπινη και εκτιμητρική χρήση και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Γιούσο, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και πάλι το δεύτερο ηλεκτρονικά, συμβασμός για την πρόταση περί κτηνιατρικών φαρμάκων. Είχαμε ένα πολύ μικρό σκύλο φάκελο. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Πλήρης υποστήριξη. Συγχαρητήρια, κυρία Γκροστέτ. Και σε όλους όσους ε, συμμετείχατε σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Τώρα, Ψηφίζουμε την ερώτηση στην Κομισιόν για τη διάσκεψη των Ηνωμένων για την αλλαγή του κλίματος ε, στο Κατοβίτσε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη, εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει ερώτηση στο Συμβούλιο για προφορική απάντηση, με έτοιμο προφορική απάντηση, ε, προφορικής απάντησης για το Κατοβίτσα, έρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε στην ερώτηση με την προφορική απάντηση για την Κομισιόν, για την Όσο Λάιμ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Και πάλι ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την ε, ερώτηση με την προφορική απάντηση στην Κομισιόν για το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία, άρχη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Το ίδιο. Ερώτηση με έτοιμη προφορική απάντηση ε, προ το Συμβούλιο για την κυκλική οικονομία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την ερώτηση με τη μορφωφορική απάντηση ε, που απευθύνεται στην Κομισιόν. Χρήση κάναβη για φαρμακευτικού σκοπού. Άρχεται η ψηφοφορία. Η συνάδελφη εδώ προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος, αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού, για την άκετα πρίδη, για χρήση σε βιοκτώνα του προϊόντων 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Και απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε για τον προπολογισμό του 2019, εντολή για τον τριμήρη διάλογο. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την εφαρμογή τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, Επιλογέ σχετικά με θέματα διαπαφή μεταξύ τη νομοθεσία για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα. Με ανατασή χειρό. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ είναι υπέρ κατά. Κατά. Να ελέγξουμε. Γιατί μπερδεύτηκα άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη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 αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ 26 Συγγνώμη, 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά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 Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Μπορείς να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για να το ξανακάνουμε, αλλά δεν σηκώσατε τα χέρια σας. 65, ποιος είναι υπέρ. Όλοι είναι υπέρ, εγκρίνεται. Αλλά αν δεν ε, κάνετε ένα τεσσιχυρός, σύμβαστε και δύο υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την 71 άρχεται η ψηφοφορία λήξη εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ για να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάουτ, 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 77 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά. Φιλελεύθερη υπέρ κατά. Υπέρ εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Και εγκρίνεται. Ομόφωνα. Ας προχωρήσουμε το επόμενο θέμα, τη διτή ιδιότητα προϊόντων στην ενιαία αγορά. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Ναι. Έχετε ζητήσει καταρνήματα ψηφοφορία εντός του ΕΛ και ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. And it's closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές 62 διορθώνουν την πρόεδρο. Τι είπα, 62 είπα. Α, ζήτω, συγγνώμη, την 62 κοίταζα. Ναι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13α υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 13α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13β υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. And it's closed and it's adopted nearly. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται από σχεδόν όλους. Ε, τροπολογία 102. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Compromise 15 in Ε, συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, η ηλεκτρονική επαλήθευση της 15. The vote is open and now it's closed. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 130 με προφορική τροπολογία. Μάλλον, ε, καταρχάς, υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 130 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 με προφορική τροπολογία πάλι, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ψηφίζουμε την 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές. Το ΕΛΚ στη 46 τι ψηφίζει. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται. 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία. What is she doing there? Can you see And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. There a lot of Ψηφίζουμε τώρα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ε, κατά της μικροβιακής αντοχής. Συμβαστική τροπολογία 1. Α, όχι, συγγνώμη. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Τροπολογία 80. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, άποχε, εγκρίνεται. Πρώτη συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. δύο κατά 96 υπέρ, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έλεγχος για το 91. Ψηφίζουμε για το 91. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Πάμε στο 96 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 96. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 99. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 κατά αποχές εγκρίνεται. 45 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ταυτόσιμη 125, 126, 146. Και παρακάτω, όχι, όχι, όχι, είναι χωριστά. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των τριών. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 128 147-130 ταυτόσιμες που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωρούμε. 143 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για το 143. Πέρας. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Απογείες απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά έλεγχος για το 152 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 12 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε όχι. 169 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά 166 υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 θεώρησε το τελμιδίο όπως πριν αλλά να ξανακάνουμε με έλεγχο την 170 και ψηφίζουμε Α, όλοι. Όμονον, καλά. Πέρασε. Ναι, και εγκρίνεται. Κατά 71, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 30 υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται. Άγκρι 10 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 8 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ συμβαστική. Εγκρίνεται. 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά απόχε, εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ. Α, όχι, το είπαμε, το είπαμε. 265 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 266 τμήμα. Σε δεύτερο τμήμα, συγγνώμη, πρώτο, εγκρίνεται άγκρι 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, α, 285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, για να είμαστε βέβαιοι. Τελικά εγκρίνεται 286 υπέρ κατά. Ε, το ελκτή είναι υπέρ κατά. Συγγνώμη, το ξανακάνουμε. 286 υπέρ κατά. Αποχές. Α, ε, σαφώς 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Το 298 ψηφίζουμε. and it is adopted. 299 in favor. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 303, υπέρ. Κατά. Αποχές, να ελέγξουμε την 303 άρχιτη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 309 και 310 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνονται. 311 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 313-314 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 315 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 317 υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία.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 κατά εποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 329 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 330 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 331 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ, κατά. Έλεγχος για την 333, άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 335 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 336 υπέρ κατά άλντε υπέρ εγκρίνεται 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγκρ 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 354 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 355 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. 356 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 370 και 371 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 393 υπέρ Κατά. Αποχές. Το άλλο είναι κατά. Απορρίπτεται. 394 υπέρ. Θέλετε ελεγχό, μάλιστα. Να ελέγξουμε την 393. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 394 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 395 και 443 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 408 να ελέγξουμε την 407 Άρχεται η ψηφορία, λήξη, εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. 408 και άγκρι 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Συγγνώμη, είμαι πολύ κουρασμένη. Κυρία Καμπεσόν, ίσως είναι λίγο αργά, αλλά έχω μια αμφιβολία. Όταν κάναμε Όταν ε, κάναμε τον έλεγχο της 393 δεν είδαμε το αποτέλεσμα γιατί δεν βγήκε στην οθόνη. 25 προς 36. Άγκρι 39, υπέρ. 408 και άγκρι 39, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 409, 410, 412, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 421 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 424 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 425 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 26 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τώρα θα το ελέγχω από εδώ και πέρα είναι μισό-μισό. Λήξη. Εγκρίνεται. Άγκρι 48 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την άγκρι 48. Εγκρίνεται λοιπόν. 4,51 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ. Κατά. Να αλλάξουμε την τέσσερα. Αφού δεν σηκώνετε τα χέρια σας, δεν ξέρω. Λήξη. Εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ. Κατά. Κοιτάξτε, βλέπω μόνο δύο χέρια. Δεν ξέρω αν είναι όλη η ομάδα. Ελέξουμε την 5. Άρχιε η ψηφοφορία. And Λήξη. Συγγνώμη, αλλά δεν είδα τα χέρια σας. Δεν κάνατε ένα τεσχυρός. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 7 υπέρ κατά Αποχέ συγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 11 και 12 υπέρ κατά αποχές συγκρίνονται. 13 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά έλεγχος. Άρχεται η σοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 15, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει, 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να επιστρέψουμε στη 16, μάλιστα βεβαίως, να ελέγξουμε τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Εντάξει, όταν είναι πολύ κοντά το αποτέλεσμα θα ελέγχω. Πού είχαμε μείνει, 22. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 και 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 35 άρχεται η ψηφοφορία λήξη απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε Άρχεται η ψηφοφορία για την 36. And Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά ελέγχου ελέγχουμε τη 46 έρχεται ψηφοφορία λήξη εγκρίνεται 47 υπέρ είπα ότι εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά εποχές εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροφολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά μπορούμε και να το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Λήξη. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 63 κατά 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά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 3, συγγνώμη, 71 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά. αποχέ, απορρίπτεται. Αν θέλετε μπορούμε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 73, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την 74 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Ήτρε B, β, υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. Ήτρε C, υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. Ήτρε D, υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Ήτρε ή ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε I, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε M, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77, υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 77, άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται 78 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Ήτρε κάπα υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και ζητώ συγγνώμη από την κυρία Καμπεσόν. Ε, τα λάθη που έκανα πραγματικά δεν ήταν ηθελημένα. Έτσι κλείνουμε τις ψηφοφορίες και περάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Σας δίνω δύο λεπτά να εγκαταλείψετε την αίθουσα αν το θέλετε. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους που συζητούν εντός της αιθούσης να συνεχίσουν τη συζήτηση εκτός της αίθουσας. Ελκ, σας παρακαλώ. Hello. Could you continue possibly outside the room? Μήπως θα μπορούσατε παρακαλώ να συνεχίσετε τη συζήτηση εκτός της αιθούσης. Και συνεχίζουμε κατευθείαν με το σημείο 20 της ημερησίας διάταξης, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμονους οργανικούς ρήπους. Αναδιατύπωση, η συγγήτρια είναι η Julie Γκέρλινγκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για απλή αναδιατύπωση. Αν μπορεί κανείς ποτέ να θεωρήσει μια αναδιατύπωση απλή Στόχος είναι η ισχύουσα νομοθεσία να ευθυγραμμιστεί με την επικαιροποιημένη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμονους οργανικούς ρήπους. Κάτι που γίνεται περιοδικά. Όπως λέει ο τίτλος, η έμονη οργανική ρήπη, POP στα αγγλικά, είναι ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον για πολύ, χρονικό, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από την αρχική τους χρήση. Πολλοί από αυτούς ε, αρχικά ήταν φυτοφάρμακα ή βιομηχανικά χημικά που μπορεί κατόπιν να εισέλθουν στην ε, τροφική αλυσίδα και έχουν ε, σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Πρόκειται για έναν από τους τομείς όπου έχουν γίνει πολλές πρόσφατες έρευνες και στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να μετράμε, αλλά ε, οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας. Ιδιαίτερα λοιπόν όσον αφορά τη συγκέντρωση των έμονων οργανικών ρήπων στη Μεσόγειο, στην ε, Βόρεια Ακτική θάλασσα και την Ανταρκτική. Ε, επικαιροποιούνται συνεχώς με νέα δεδομένα. Από τότε που ανακαλύψαμε τις ιδιότητες των έμονων οργανικών ρήπων, η χρήση τους απαγορεύτηκε με μόνο κάποιες ελάχιστες και πολύ αυστηρές παρεκκλήσεις. Με τη σύμβαση της Στοκχόλμης, τη διεθνή αυτή σύμβαση, Πιστεύουμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Ο εντοπισμός νέων χημικών ουσιών και η συμπερίληψή του στην ομοθέσια συνεχίζεται κανονικά ε, σε διεθνές επίπεδο. Τι έκανα εγώ λοιπόν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι αρκετά απλή και σαφής αναγνωρίζει νέο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, κάτι που νομίζω ότι θα επικροτήσουν οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ. Έχω υποβάλει κάποιε τροπολογίε που στόχο έχουν να ενισχύσουν το νέο αυτό ρόλο ε, του οργανισμού. Έχω συνομιλήσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σχετικά με τον νέο ρόλο. Υπάρχουν κάποια θέματα δημοσιονομικά, αλλά γενικά ο οργανισμός ε, χαιρετίζει αυτόν τον νέο ρόλο που του δίδεται. Φαίνεται λογικό να αναλάβει τις εργασίες αυτές, τα καθήκοντα αυτά ο ΕΚΑ. Πρέπει να θίξω ένα θέμα που με ανησυχεί, που είναι η έλλειψη μελέτης αντικτύπου. Επειδή πρόκειται για απλή αναδιατύπωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι αυστηρά απαραίτητη μια μελέτη αντικτύπου, κάτι που μάλλον θα μας πει κιόλας τώρα που θα πάρει το λόγο. Δεν συμφωνώ με το θέμα αυτό όμως, διότι ακόμα και σε περίπτωση αναδιατύπωσης ε, θα πρέπει να έχουμε μια μελέτη αντικτύπου. Θα περιμένω να ακούσω τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Γνωρίζω καλά τη, τη χρονική πίεση, θα ήταν θετικό να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό μέχρι το τέλος της θητείας μας. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας οι σκιώδεις εισηγητές κατά τη διάρκεια της πρώτης μας ε, συνάντησης, πόσο μάλλον που δεν έχουμε την μελέτη αντικτύπου. Διότι στις συζητήσεις που είχαμε με διάφορους ενδιαφερομένους, και ιδιαίτερα στην περίπτωση κάποιων από αυτά τα προϊόντα με ανθρώπους από τον βιομηχανικό κλάδο, θεωρούν ότι υπάρχουν επιπτώσεις περιβαλλοντικές και εμπορικές που θα έπρεπε να αξιολογηθούν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Κάποιες τροπολογίες δικές μου προσθέτουν κάποιες ουσίες στα παραρτήματα και οι σκιώδεις μάλλον θα έχουν αναρωτηθεί από πού προέκυψαν οι ουσίες αυτές. Μου ζητήθηκε να συμπεριλάβω τις ουσίες αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόλαβε την προθεσμία για τις ενδοϊπηρεσιακές διαβουλεύσεις της. Ευχαρίστως λοιπόν συμπεριέλαβα ε, τις ε, ουσίες αυτές, ε, παρότι τις έλαβα τελευταία στιγμή. Μετά την δημοσίευση των τροπολογιών μου, είχα πολλές επαφές, ιδιαίτερα όσον αφορά το δεκαβρομοδιφενήλεθέρα, διότι Καθορίζεται εδώ ένα όριο το οποίο δεν υπάρχει στη σύμβαση της Στοκχόλμης. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και ενδεχομένω να ε, κάνουμε και κάποιες αλλαγές ακόμα. Υπάρχουν κάποιες συνέπειες ιδιαίτερα για την ανακύκλωση και από ό,τι καταλαβαίνω το θέμα αυτό συζητιέται και στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας για την ανακύκλωση αποβλήτων. Ε, πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε τις διάφορες αυτές διαδικασίες. Γνωρίζω λοιπόν ότι μάλλον απαιτεί περισσότερη εξέταση το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει σε διάφορα κράτη-μέλη, όχι όλα, έχει να κάνει με την ε, χρήση των PCB ε, στα ε, εθνικά ηλεκτρικά δίκτυα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει προθεσμία για την κατάργηση της χρήσης των πολυχλωριωμένων διφενηλίων. Ε, αυτό δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Ε, πάντα θεωρείται ότι η τροποποιήσεις αυτές ε, θα γινόντουσαν ε, με ανανέωση του εξοπλισμού. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις συνέπειες. Όταν λέω ότι το θέμα αυτό προκύπτει σε κάποια κράτη-μέλη, ε, το ανησυχητικό είναι ότι πολλά δεν γνωρίζουν πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα PCB, τα τη φενήλια, στα ηλεκτρικά τους δίκτυα. και χωρίς ε, να θέλω να υπονοήσω ότι ε, μπορεί να μην ε, γίνεται σοφή χρήση, νομίζω ότι είναι ανησυχητικό ότι δεν γνωρίζουμε στοιχεία ακριβή για την χρήση αυτών των ουσιών. Όπως σας είπα λοιπόν, πρόκειται για σχετικά απλή πρόταση. Ε, δεν είχαμε ακόμα ε, ενελεχή συζήτηση με του κοιόδης εισηγητέ. Ελπίζω όμω να μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ, Τζούλη. Οι εισηγητέ ε, τώρα. Ε, δίνω το λόγο στον Μάσιμο Παουλίουτσι. Ναι, ευχαριστούμε για τη δουλειά σα. Τώρα έχουμε αυτέ τι τροπολογίε 3, 4 και 12. Ε, ήμουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το κύμα της Στοχόλμης. Πρέπει να ακούσουμε βέβαια επί της την άποψη της ε, Κομισιόν. Και έχουμε και εμείς κάποιες τροπολογίες. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε τις διατάξεις για το πώς πώς θα προστατευτεί η υγεία, πώς θα υπάρχει περισσότερη ενημέρωση του κοινού. Τώρα, όσον αφορά τους ε, τόπους που έχουν ρηπανθεί, θα πρέπει να αναπτυχθεί στρατηγική για αυτές τις ουσίες πόψη. Όμως, έχουμε τον κανονισμό για τον υδράργυρο, οπότε θα πρέπει να συνεργαστεί η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη για να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τους τόπου που έχουν αυτέ οι βλαβερές επικίνδυνες ουσίε. Επαόριστον λοιπόν καθορίστηκε να γίνει η αναθεώρηση του κειμένου με συνεργασία του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Για το ECR τώρα, ο επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, έχω μελετήσει το κείμενο πρόσφατα και δεν έχω να πω και πολλά στον αυτές τις λεπτομέρειες το ECR θεωρεί θετική την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για τη δουλειά της ιδίως για τροπολογίες 2 και 4. Αυτές που είναι στο και του σχήματος με τον κανονισμό Ρίτσα. Δεν έχω ειδικέ γνώσει στο θέμα, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Πρώτα πρώτα, έχουμε τώρα τους νέους κανόνες που θεσπίζουν υποχρεώσεις για την ε, υπηρεσία χημικών προϊόντων. Οπότε και η υπηρεσία αυτή θα διαχειριστεί τι υποχρέωσει που απαραίουν από αυτόν τον κανονισμό και θα εξασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία του κανονισμού από αυτή την υπηρεσία. Θα υπάρχει επρικοδότηση για αυτή την υπηρεσία, την ΕΚΑ. Δεν ξέρω θα, ε, τι θα γίνει να ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει κάποια αναβάθμιση ενίσχυση της υπηρεσίας επίση, Κάποια κρατημέλια επικρίθηκαν, για, επέκριναν μόνο την Επιτροπή για κάποιες διαδικασίες DDK και DDA αυτές οι ουσίες που έχουν κάπως ε, ανελαστική ρύθμιση σε σχέση με το αν είναι έφλεκτες και βλέπουμε εδώ τους περιορισμούς όσον αφορά την ευθυγράμμιση REACH και κειμένου στο χώρο μας. Η στόχη είναι διαφορετική. Οπότε και εμείς προβληματιζόμαστε μια που δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ξεκάθαρες προβλημόνες διαδικασίες. Φερρυπίν όσον αφορά τις οριακές τιμές. Τι γίνεται, πώς εντάσσεται αυτό στην κυκλική οικονομία. Δεν θα πρέπει η Κομισιόν να τα κάνει τα πράγματα πιο διαφανεί. Πάντως θα συνεργαστούμε τις άλλες πολιτικές ομάδες για το θέμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την συνένεση και συμφωνία με το Συμβούλιο κατά αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Άλντε. Ο ο κύριος συνάδελφος, ποιος είναι. Κύριος Μπέντερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ καλή δουλειά τη συναδέλφου. Ελπίζουμε θα ολοκληρωθεί σύντομα το θέμα. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και εγώ θεωρώ πως είναι σημαντικό το τώρα η καινούργια υπηρεσία για τα χημικά έχει εμπλακεί. Μία ερώτηση όπως την Επιτροπή. Τα κράτη με λένε ότι δεν είναι σαφές το πώς γίνεται ο ορισμός, καθορισμός των ΠΟΠ καμιά φορά όμω ε, πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη και δεν είναι εντύπωση ότι για το αίτημά του τίποτα δεν έχει γίνει. Μήπω θα πρέπει να είναι με μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο ανοιχτή, πιο ξεκάθαρη όσον αφορά τα απόψη. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, κυρία Κονίτσνα, για την Γκουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ Τζούλη για όλο σου το έργο και μερικές φορές ε, λεπτομερείς ε, τροπολογίες ε, θεωρούνται ότι είναι εντάξει αλλά να έρχονται από την Κομισιόν, καλό είναι να το ξέρουμε. Επίσης, όπως είπε, ευθυγρασμός εδώ με τη ε, σύμβαση της Στοκχόλμη ε, και έχουμε την DKBD που υπάρχει εδώ και χρόνια. Είναι καλό που γίνεται αυτή η ευθυγράμμιση, γιατί είναι σημαντικό γιατί ε, θα πρέπει να βγει εκτός του συστήματος, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολλά ε, πολλές ουσίες ε, μέσα, πρέπει να ξέρουμε όταν ανακυκλώνουμε ότι έχουμε και οριακές ε, τιμές. Έτσι λοιπόν, σας υποστηρίζω εδώ. Όμως έχω ένα μεγάλο ερώτημα και ερώτηση για την τροπολογία 12, γιατί έχουμε και πάλι μια τετρασέλιδη τροπολογία. Θέλω να ρωτήσω και αυτή είναι από την Κομισιόν. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό είναι τι κάνει ακριβώς η συγγήτρια εδώ. Λέει ότι για λόγους καλύτερης νομοθεσίας. Όταν λέει κάτι τέτοιο, εγώ το διαβάζω πιο προσεκτικά. Τι ζητάμε. Ο Οργανισμός Χημικών Ουσιών να εξετάσει αν είναι μόνος οργανικός ρήπος μία ουσία, ναι ή όχι, αλλά να το κάνει αυτό ε, ε, χρειάζεται να αξιολογηθεί ένα τεράστιο κατάλογος οικονομικών και κοινωνικών δικτών. Εγώ δεν νομίζω ότι για τον προσδιορισμό ε, ή για το αν είναι δηλαδή μία ουσία μόνος οργανικός ρήπο ή όχι, πρέπει να κάνει κοινωνικο-οικονομική ανάλυση. Το κάνει μετά. Αν έχει προσδιοριστεί ω pop, μπορεί να το αλλά για την ταυτοποίηση ως οργανικός ρήπος λοιπόν, δεν χρειάζεται να μπαίνει σε οικονομικές ε, περιστάσεις και θέλω να μου πει η Κομισιόν περί τίνος πρόκειται γιατί έχουμε δύο σελίδες και λέει ότι πρέπει να δούμε την ε, ε, τεχνική δυνατότητα, ε, τα οικονομικά στοιχεία. Εδώ προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τους όμορους οργανικούς ρήπους. δεν καταλαβαίνω όλα αυτά περί διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της αξιολόγησης, γιατί τα μπερδεύουμε εδώ αυτά και κατά τη δική μου άποψη αυτός δεν είναι ένας καλός κανονισμός. Έτσι λοιπόν, άμεση ερώτηση των Κομισιών, τι πιστεύει γι' αυτό, για αυτή τη διεύρυνση Τη της εισηγήτριας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ελπίζω να είναι η σειρά για την ε, εισηγητρία της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Ε, ε, Συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την Τζούλη Κέρλινγκ για την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσής της. Επικροτώ την έκθεση αυτή διότι αποτελεί απαραίτητο βήμα για την εφαρμογή των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις. Έχουμε λάβει πολύ πρόσφατα το έγγραφο αυτό, έπρεπε να το έχουμε εδώ και αρκετό καιρό και έχουμε καθυστερήσει κάπως. Ε, δεν φταίει όμως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα παραρτήματα ε, θα τροποποιούνται με κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτό δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Επίσης, εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επίτροπης ε, για έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Ούτε και αυτό το βρίσκω σωστό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, να μπορεί τουλάχιστον να απορρίψει τις σχετικές προτάσεις. Τρίτον, δεν ε, μου αρέσει η παρέκκληση ε, για τις παραφίνες. Ε, τέταρτον, είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να ασχοληθούμε και με τα απόβλητα και την ανακύκλωσή τους. Πιστεύω ότι είναι ανεπαρκής η ρύθμιση για τους έμονους οργανικούς ρήπους, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει μεν κάποιες οριακές τιμές για τον δεκαβρομοδιφενήλεθέρα στις ε, οικοδομές, ε, αλλά θα πρέπει να έχουμε οριακές ε, τιμές ε, και στα απόβλητα. Επιπλέον δεν θα πρέπει να έχουμε τόσες παρεκκλήσεις για έμονους οργανικούς ρήπους σε άλλα προϊόντα. Κάποια κράτη-μέλη δεν τηρούν τις ε, διατάξεις αυτές όπως απαιτεί και η Σύμβαση της Στοκχόλμης. δεν ε, πληρούνται όλες οι απαιτήσει ε, της σύμβαση της Στοκχόλμης. Όσον αφορά τις ε, διαβουλεύσεις με τον τομέα αυτών, περιορίζεται ο ρόλος των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών μας πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα. Θα υποβάλουμε τροπολογίες. Τζούλη, προσλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει η Κομισιόν. Παρακαλώ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, κ. Στόπικ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέρλινγκ για το σχέδιο έκθεσης και για όλα τα σχόλια που κάνατε για το σχέδιο έκθεσης και για την πρότασή μας. Όπως ήδη υπόθηκε από την εισηγήτρια, ο κανονισμός των έμονων οργανικών ρήπων έχει θετηθεί το 2004 και εφαρμόζει την ε, συνθήκη της ε, Στοκόλμης για τους έμονους οργανικούς ρήπους που επίσης ε, τέθηκε σε ισχύ το 2004. Η σύμβαση της Στοκόλμης είναι μια παγκόσμια συνθήκη ε, υπό τον ΟΗΕ και ρυθμίζει τους έμονους οργανικούς ρήπους ε, παγκόσμιας ανησυχίας. Η συγγήτρια εξήγησε ήδη ότι οι έμονοι οργανικοί ρήποι μένουν στο περιβάλλον για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, είναι πάρα πολύ τοξικοί, ταξιδεύουν γύρω από τον πλανήτη και αποτελούν απειλή για όλους ε, που ζουν στον πλανήτη και τους ανθρώπους, αλλά και όλα τα ζώα και τους ζωντανούς οργανισμούς εν γέννη. Επομένως, είχαμε τις διαπραγματεύσεις και την οριστική έγκριση και θέση εφαρμογή της σύμβασης αυτής, προκειμένου να ρυθμίσουμε τους όμως οργανισμούς ρήπους παγκοσμίω. Ο κανονισμός των ΠΟΠ εφαρμόζει τη συνθήκη της σύμβαση της Στοκχόλμης και μεταφέρει όλες τις υποχρεώσεις των μερών σε νοσιακό δίκαιο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εντός της Ένωσης υπάρχει ένα ρεμονισμένη νομοθεσία που αντιμετωπίζει ε, αυτούς ε, τους οργανικούς ρήπους λοιπόν, αναθεώρηση, αναδιατύπωση του κανονισμού ΠΟΠ. πυροδοτήθηκε από την ανάγκη ευθυγράμμιση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων με τη Συνδίκη τη Λισαβόνα. Αυτό είναι ο κύριο στόχο αυτή τη σύμβαση. Επομένω, προτείνουμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε κατεξοδότηση πράξη και εκτελεστικές πράξεις ε, όπου δει. Επιπρόσθετα, δίνουμε στον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ένα ρόλο, καθώς ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων είναι ο κύριος κόμβος για επιστημονική και τεχνική γνώση στην Ένωση για θέματα χημικών. Και αυτός ο κανονισμός και η σύμβαση απαιτούν επιστημονική συνεισφορά και τεχνική συνεισφορά και φυσικά όλοι ωφελούνται ε, με την εμπλοκή του ΕΚΑ και δημιουργώντας και συνέργειες με όλη την άλλη δουλειά που κάνει η ΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, προτείνουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, για τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης σύμφωνα με την, το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία και σύμφωνα με τον ελέγχο κατανότητα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε καλύτερη ενημέρωση του κοινού στα κρατη και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη υποβολή εκθέσεων προς την Σύμβαση της Στοκόλμης. Επίσης, επικαιροποιούμε κάποιους ορισμούς για να τους ευθυγραμμίσουμε με πιο πρόσφατες νομικές πράξεις όπως το ΡΙΤΣ. Επομένως, ο κύριος στόχος αυτού του κανονισμού είναι η εφαρμογή της σύμβασης και ο κύριος στόχος της σύμβασης είναι η εξάλληψη των έμονων οργανικών ρήπων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Νομίζω ότι αυτά όλα θα πρέπει να τα, όλοι θα πρέπει να τα έχουν κατά νου όταν εξετάζουν αυτή την πρόταση. Η συγγήτρια ανέφερε την ε, έλλειψη μελέτης αντικτύπου. Όπω είπαμε στην πρότασή μα, δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη μελέτη αντικτύπου, γιατί δεν τροποποιούμε στην πραγματικότητα τον κανονισμό αυτό. Ούτε τη λειτουργία του κανονισμού, ούτε τι υποχρεώσει που έχουν τα κράτη-μέλη ή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επομένως, δεν θεωρήσαμε ότι υπήρχε ανάγκη για μελέτη αντικτύπου. Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις για την εμπλοκή του οργανισμού χημικών προϊόντων και τον προπολογισμό. Από δημοσιονομική σκοπιά πιστεύουμε ότι η πρότασή μα. λαμβάνει υπόψη το αναμενόμενο άχθος εργασία ε, για τον ΕΚΑ, γιατί ξέρουμε τι αναμένουμε από τον ΕΚΑ στο μέλλον, όπως είπε και η συγχύτρια, εμείς ε, αναθέτουμε και συμβάσεις ε, σε εξωτερικούς συμβασικούς που μας δίνουν επιστημονική και τεχνική βοήθεια. Αυτό το έργο τώρα θα γίνεται από τον ΕΚΑ, αλλά ΕΚΑ θα κάνει περισσότερα από αυτούς ε, τους υπεργολάβους και αυτό δεν κατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό μας. Τώρα, στρέφομαι σε ορισμένε πιο συγκεκριμένε ερωτήσει που τέθηκαν. να ξεκινήσω με τις ε, κοινωνικο-οικονομικές πτυχές ε, και την τροπολογία 12 και το μικρή κατάλογο κριτηρίων. Όπως βλέπετε στην πρότασή μας, εμείς δεν έχουμε προτείνει ένα τέτοιο κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε ένα φάκελο που θα καλείται να προετοιμάσει ο οργανισμός χημικών προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία προσδιορισμού των νέων ΠΟΠ. Δεν υπάρχει υποχρέωση δυνάμει τη σύμβαση του κανονισμού για τον προσδιορισμό νέων αίμονων οργανικών ρήπων. Αυτό είναι στα μέρη να αποφασίσουν αν ε, θέλουν να προσδιορίσουν ε, νέους οργανικούς ρήπους. Όμως ενθαρρύνονται τα μέρη να επενδύσουν ε, στον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων ΠΟΠ που θα υποβληθούν στη συνέχεια στη διαδικασία που περιγράφεται στη σύμβαση. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μια αναθεώρηση που θα γίνει από την Επιτροπή Αναθεώρησης των ΠΟΠ στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν 31 εμπειρογνώμονε που διορίζονται από τα μέρη. Οι εμπειρογνώμονε αυτοί εξετάζουν τι προτάσει που καταθέτουν τα μέρη. Και η πρόταση ενό μέρου ε, ζητάται να συνοδεύεται από ένα φάκελο, ο οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίε σύμφωνα με το παράρτημα Δέλτα τη ε, σύμβαση, στα κριτήρια ελέγχου. Αυτά τα κριτήρια υπάρχουν προκειμένου να προσδιορίσουμε αν ε, μια χημική ουσία πληρεί τα κριτήρια POP ή όχι. Και υπόθηκε σε κάποια παρέμβαση ότι ο προσδιορισμός ταυτοποίηση ενός POP δεν ε, έχει κοινωνικο-οικονομικές πτυχές. Γίνεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων και αυτά τα κριτήρια αφορούν τις ιδιότητες ε, της χημικής ουσίας. Η ερώτηση είναι αν μια χημική ουσία έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. και αυτέ οι ιδιότητε περιγράφονται στην ε, Σύμβαση της Στοκχόλμης. Έτσι λοιπόν, υπάρχει στη Σύμβαση ένας κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται μαζί με την πρόταση και που πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή Αναθεώρηση ΠΟΠ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Εξέτασης ε, ελέγχει τα κριτήρια αυτά και καταλήγει στο συμπέρασμα, αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια πληρούνται για μια χημική ουσία, πάμε στο επόμενο βήμα, το ε, προφίλ κινδύνου, risk profile, που καθορίζεται από την Επιτροπή για τους πόπες, συλλέγονται όλες οι πληροφορίες για το χημικό αυτό και για τους κινδύνους που εμπλέκονται στη χρήση του χημικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση από όλα τα μέρη παγκοσμίω και οι κινδύνοι που μπορεί να προκύψουν. Και στη συνέχεια η Επιτροπή Εξέτασης προβαίνει σε μια αξιολόγηση διαχείρισης του κινδύνου σε αυτό το βήμα εξετάζουν ε, λεπτομερώς ε, τις χρήσεις, τις εναλλακτικέ και εκεί λαμβάνεται υπόψη και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές. Εκεί θα πρέπει να εξεταστούν οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και πληροφορίες. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό στο στάδιο του προσδιορισμού, του δορισμού, γιατί αυτό απαιτεί μόνο επιστημονικά κριτήρια. Και υπήρχε για μια ερώτηση αν τα κρατημέλη μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση. Πράγματι μπορούν. Και ήδη έχουμε μια πολύ εύρωστη διαδικασία, γιατί βράζουμε τα δυνατά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη έχουμε μια συνάντηση ερμηδιών αρχών για το ΠΟΠ, όπου τα κράτη-μέλη και κομισιόν συζητούν και για τον προσδιορισμό νέων ΠΟΠ. Ε, έχουμε ε, φακέλους που κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών για σχολιασμό και έχουμε μπλέξει και τον ΕΚΑ ως ένα βαθμό. Δεν έχει ο ΕΚΑ εντολή, όμως ε, έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το PBT ε, και μας ε, Συμβουλεύουν οι εμπερογνώμονε για τα κριτήρια PBT που είναι κοντά στα κριτήρια POP. Έτσι λοιπόν υπάρχει ήδη μια βρωστή διαδικασία στην Ένωση και δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια διαδικασία προσδιορισμού να περιγράφεται στον κανονισμό. Αυτό περιγράφεται και από την απουσία τέτοια διαδικασία ε, προσδιορισμού στην πρότασή μα. Και τώρα, Πρόεδρε, να αναφερθώ στα τελευταία σημεία που αναφέρθηκαν από τους βουλευτές, ε, το θέμα της κατηγοριοποίησης του DKBD. Η, σύμβαση, η διάσκεψη των μερών το 2010 αποφάσισε για τα πολυχλωριωμένα διφενήλια ε, τέτρα, πέτρα, πέντα και έξα και η απόφαση αυτή ελήφθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο για να υπάρχει εξαίρεση ανακύκλωσης προϊόντων που περιλαμβάνουν, που περιέχουν αυτά τα χημικά προκειμένου να επιτραπεί ένα βαθμό η ανακύκλωση, αντικατοπτρίζεται αυτή η εξαίρεση και στο παράρτημα του κανονισμού που που αναφέρονται αυτά τα PBDs και το έξα ε, προμοντάιν αναφέρθηκε ε, από τη διάσκεψη των μερών, δεν έχει αντικατοπιστεί ακόμα στην πρότασή μας λόγω χρονοδιαγράμματος. Αυτή η απόφαση λήφθη σε διεθνές επίπεδο και δεν περιλαμβάνει εξαίρεση ανακύκλωσης. Δεν έχουμε λοιπόν εξαίρεση ανακύκλωσης για τον 10 προμοντάιλ φενίλ ε, υπάρχει περιορισμός για τη χρήση του DKBD στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει εξαίρεση για την ανακύκλωση. Επομένως, το κείμενο όπως έχει παρουσιαστεί στην έκθεση της εισηγήτριας δεν ε, αναφέρεται σε κάποια εξαίρεση ανακύκλωσης ε, που δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το σχέδιο κειμένου είπε συγκέντρα ότι προτείναμε αυτό το κείμενο. Είναι σωστό να προτείνουμε κείμενο στην εισηγήτρια, καθώς μας ζητήθηκε να παράσχουμε μια πρόταση. Και το κείμενο αυτό παρουσιάζει τα διαθέσιμα στοιχεία, την απόφαση που λήφθη από τη διάσκεψη των μερών, τον περιορισμό που έχει διευθυνθεί υπό το ΡΙΤΣ και την εντολή που πήρε η Κομισιόν από το Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί στη διάσκεψη των μερών. Καθώ, όπω ξέρετε, κάθε διάσκεψη των μερών, σε ό,τι αφορά τι αποφάσει κατηγοροποίηση, καταλογοποίηση, χρειάζεται μία εντολή και βάσει τη εντολή διαπραγματεύεται η Κομισιόν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και αυτά περιλαμβάνονται στην πρόταση για την καταλογοποίηση του DKBD. Σας ευχαριστούμε για τη λεπτομερή εξήγηση. Ελπίζουμε ότι η Κομισιόν πάντοτε θα μας δίνει τόσο λεπτομέρειες εξηγήσεις. Ε, Τζούλη, θες να προσθέσεις κάτι. Είσαι γύτρια. Σας θα πω ανάποδα, ίσως από το τελευταίο. Τα είπα λεπτομέρως, όχι πολύ λεπτομέρως. Γιατί υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Κυρίως για τις τιμές. Οπότε να συνεργαστούμε με τους και την ε, Κομισιόν όταν συναντηθούμε. Τεχνικό είναι το θέμα, αλλά σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το νέο μου παράρτημα. Ε, βέβαια, και έτσι θα ευθυγραμμίσουμε το κείμενο με το REACH. Το συζητήσουμε. Ναι τον συνάδελφο και όσον αφορά τις ε, οικονομικές προ προς την υπηρεσία χημικών από ό,τι ξέρω μετά τη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή έχει προταθεί να γίνει πρόβλημα στον προπολογισμό για τέτοια προϋποδότηση και ο Γενικός είναι ικανοποιημένος, οπότε δεν το αμφισβητώ. Επομένως, ναι, σας διαβεβαιώ, υπάρχει πρόβλεψη. Α, και κάτι άλλο για τον κύριο Παολούτσι. Για αυτά τα μολυσμένα μέρη. Θα το δούμε. Δεν το σκέφτηκα. Δεν το συζητήσαμε τους κοιόδες, αλλά είμαι ανοιχτή σε προτάσεις να το συζητήσουμε. Στην πρώτη μας συνάντηση με τους κοιόδες θα το πούμε, θα το κανονίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η 27 Ιουνίου στις 11 η ώρα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Στην ΕΝΒΗ θα ψηφίσουμε 10 Οκτώβριο. Στην Ολομέλεια, α, όχι, όχι. Πάμε τώρα στο 21 που είναι Η σε εγκαταστάσεις παραλαβή αποβλήτων πλοίου. Α, αυτή τη φορά δεν θα την πατήσω. Και ο κύριο Έκχαουτ θα είναι ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο. Είναι εισηγητής. Έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μα το ήθελα να πω και εγώ ότι τουλάχιστον τώρα θα πετύχετε τη σειρά. Α, εδώ πέρα σκεφτήκαμε το ίδιο. Σα και σας ευχαριστώ. Πρόκειται για κάποια γνωμοδότηση για την Τραν. Με χαρά. Βλέπω ότι είναι εδώ και ο εισηγητής ή η εισηγήτρια. Οπότε δύο σε ένα γιατί είστε και σκιώδης της ε, Άλντε. Οπότε, να, για πέστε μου πώς θα τα συνδυάσετε. Πολύ σημαντικό το θέμα. Έχει σχέση με την στρατηγία τα πλαστικά και η Κομισιόν έχει δύο προτάσεις. Ε, πρώτον η πρόταση για την ε, μία χρήση και εδώ όσον αφορά την ρήπανση της θάλασσας και τι θα γίνει με αυτό. Πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα σκουπίδια προέρχονται από την γη αλλά το 1 τρίτον προέρχεται και από τη θάλασσα. Οπότε βγαίνει ο γένος. Οπότε δεν υπάρχει κίνητρο, μάλλον αντικίνητρο υπάρχει όσον αφορά τα πλοία για να, να μαζεύουν τα απόβλητα και να τα φέρνουν στο λιμάνι, σε κάποιο λιμάνι. Πρέπει κάτι να καταβάλουν και όσο περισσότερα από όλα τα φέρουν, τόσο περισσότερο πρέπει να πληρώσουν. Ε, αυτό δεν είναι κίνητρο, ούτω ώστε κάποιο να φέρνει τα απόβλητά του στην ξηρά. Οπότε είπαμε 100% να καταργηθούν αυτά τα τέλη. Και θα υπολογίζεται πόσο κοστίζει ο πλουράς λιμένος πόσο κοστίζει στο κάθε σκάφος το να μεταφέρει τα απόβλητα. Πάντως, τα λέει και η Κομισιόν και εγώ ως εισηγητής προσπαθώ να βελτιώσω το κείμενο ότι ας πούμε όσον αφορά το, το, ένα πράσινο σκάφος θα πρέπει κανείς να αποδείξει ότι με, με οικολογικό τρόπο κανείς μεταχείριζε τα απόβλητα. Όταν λοιπόν εφαρμόζει αυτού του είδους την ε, μεταχείριση, αυτή τη διαχείριση, τότε κανείς αντί να καταβάλει το τέλος έχει έκπτωση. Να, ένα κίνητρο τόσο ώστε να υπάρχει διαχείριση των αποβλήτων ή οικολογική. Αυτό προτείνουμε. Θα γίνει ειδική συζήτηση όσον αφορά τα ληφτικά εργαλεία, όσον αφορά τα ληφτικά σκάφη, γιατί είναι πάρα πολλά τα δίχτυα τα οποία πετάγονται, χάνονται και τελικά από το τμήμα των αποβλήτων. Από να εξασφαλίσουμε ότι και αυτά θα καλυφθούν. Γιατί όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα δίχτυα άμεσα έχουν αρκετές επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Αλλά βέβαια και οικονομικά βλάπτουν τα σκάφη. Και αυτά είναι πρόβλημα. Εγώ ως συζητητής προτείνω επίσης επιτέλους να έχουμε κάποιο είδου οικονομικό κίνητρο, ούτω ώστε όταν αγοράζει κανεί κάποιο δίκτυο στο τέλο τη ζωή του να το φέρνει πίσω το άχρηστο πια δίκτυο στο λιμάνι και να μην πετάγονται στην θάλασσα με όλε τι συνέπειε για για στα δίκτυα. Να κάποια στοιχεία γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένο με την πρόταση της Κομισιόν και προσπαθώ απλώς να θωρακίσω το περιεχόμενο σε διάφορα σημεία, αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε το ότι η ποινικοποίηση του να πετάει κανείς αυτά τα απόλυτα στη θάλασσα είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει ένα ξεκίνημα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει αυτόν πλήρως να εφαρμοστεί στην Ένωση. Επίσης, ερώτηση προς την Επιτροπή. Μια που αποφάσισαν αυτές οι πλατφόρμες, ε, οι offshore πλατφόρμες, οι υπεράκτες, να δούμε κατά πόσο θα καλυφθούν. Να το δούμε, να το δούμε, να το συζητήσουμε, να θα καλυφθούν και πώς το βλέπετε. Όποτε μπορείτε να μας πείτε. Και έτσι θα βελτιωθεί η πρόταση και οι πλατφόρμες επομένως να δούμε πώς θα τις ε, ε, εντάξουμε στη ρύθμιση. Αυτά. Πρέπει να ακούσω τι έχουν να πούν οι σκιώδες ηγητές. Να είναι καλή η ονομοδότηση. Για να σας δούμε το Συμβούλιο που έχει καταλήξει σε κάποια γενική προσέγγιση και θα πρέπει να εκείνη την επαφή με το Συμβούλιο να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ισχυρή θέση. Ευχαριστούμε κύριε Σικηταλή. Ο Πρόεδρο και τώρα οι σκιώδη ο κύριο Γκαμπού. Ευχαριστώ. Πρώτον, συγχαρητήρια. Μπράβο για τη δουλειά σα, κύριε Εκχάουτ. Το σχέδιο της οδηγίας εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική κατά των αποβλήτων πλαστικών, κατά των αυτών που απορρίπτονται στη θάλασσα. Και όπως είπατε, επηρεάζουν πάρα πολύ το οικοσύστημα στην Καταλωνία και από την κλιματική αλλαγή αλλά και από τα απόβλητα έχει πληγεί η προστατευόμενη περιοχή των εκβολών του Εύρου. Εκεί, από κύριους καιρών, κάνουμε κάποιες καμπάνιες ενημέρωσης, γιατί πρόκειται για μοναδικά μέρη και οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες. Στο Τόρεντε Μπάρα και σε άλλες περιοχές έχουν γίνει πανεβάσεις από την Ένωση. Αλλά εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να κανονίσουμε το πώς με τους στόχους που θέτουμε και πετυχαίνουμε να μην χρειάζονται καμπάνιες, να είναι πιο καθαρές οι περιοχές μας από κάθε είδους απόβλητα από τα σκάφη. Να έξω τίποτα για αυτές τις ε, υπεράκτητες πλατφόρμες για την εξώση πετρελαίου. Τι γίνεται, ε, πρέπει να δούμε ακριβώς ε, πόσο συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση των αποβλήτων. Επίσης να δούμε αν θα ε, καλυφθούν εδώ και οι πλατφόρμες για την ε, εξόριξη τέλος πάντων φυσικού αερίου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί για το κόστος και για το κόστος όλων αυτών των μέτρων μπορεί να κατεβάσουμε τροπολογίες όσον αφορά τώρα. Υπάρχουν προγράμματα για τα αλήφθηκα εργαλεία εμπλέκονται και οι αλλοίς και οι εταιρείε που αναδέχονται αυτά τα παλιά ληφτικά εργαλεία. Να μελετήσουμε το τι ισχύει και τα μέτρα να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα κάθε λιμένος. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε με αγαστή συνεργασία επεξεργαζόμενοι και τις τροπολογίες. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Βέλκεν για τους σοσιαλδημοκράτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή πρόταση γνωμοδότησής του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να καταπολεμήσουμε δραστικά, να μειώσουμε δραστικά και ε, μόνιμα τις, ε, τα, τα απορρίμματα στη θάλασσα. Και αυτή η οδηγία αποτελεί ε, πολύ καλό εργαλείο για αυτό. Ακόμα και οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί από τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων στην Ανταρκτική, για παράδειγμα. Γι' αυτό είναι πολύ καλό το να θέσουμε φιλόδοξους στόχους. Είναι καλό και σημαντικό να γνωμοδοτήσουμε πάνω στην γνωμοδότηση αυτή. Ε, κοιτώ και την Γκεζίνε. Τι μέτρα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, μη ειδικά τέλη κατά 100% συμφωνώ με τον εισηγητή διότι εάν ε, τα πλοία πρέπει να πληρώνουν ε, για την παράδοση αποβλήτων ανάλογα με το βάρος δεν έχουν κίνητρο να μην τα απορρίπτουν στη θάλασσα. Επίσης βρίσκω πολύ θετικό και, σωστοτικό, και σωστό να διευρυνθούν ε, τα μέτρα για τα απόβλητα να μην απορρίπτονται στη θάλασσα και επίσης βρίσκω πολύ σωστή την προσέγγιση οι αλληλείς ε, που μαζεύουν ε, απόβλητα στη θάλασσα, απορρίμματα στη θάλασσα να μπορούν να τα εκφορτώσουν χωρίς επιπλέον κόστος. Στην ε, κάτω Σαξονία στη Γερμανία υπάρχει ένα πρόγραμμα Fishing for ε, αλλιεύοντας απορρίμματα που ε, φαίνεται να είναι πολύ καλή μέθοδος. Ε, Μία ειδική περίπτωση θα ήθελα να αναφέρω, διότι πριν αναφερθήκαμε στους έμονους οργανικούς ρήπους. Παραφίνη. Η παραφίνη είναι ένα κερί που χρησιμοποιείται και στα φάρμακα, αλλά και ως καύσιμο και ε, επιτρέπεται να απορρίπτεται ε, στην ζώνη πέρα από τα 12 μίλια, αλλά ε, δυστυχώς φτάνει πάλι στα στις ακτές. Αυτό είναι πρόβλημα και για τα πτηνά, είναι πρόβλημα και για τους τουρίστες. Για να μην απορρίπτεται λοιπόν η παραφήνη στη θάλασσα, και να καθαρίζονται σωστά οι δεξαμενές ε, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Δεν γνωρίζω όμως αν τα μέτρα που προβλέπονται αρκούν. Έχει υποβληθεί ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο όμως ε, δεν έχουμε λάβει απάντηση, παρότι έχουν περάσει έξι εβδομάδες από τη λήξη της προθεσμίας. Ε, θα χαρώ πολύ λοιπόν εάν ε, απαντηθεί το ερώτημα των Ευρωβουλευτών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αρκεί για να αποφύγουμε Αρκούν τα μέτρα που έχουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραφήνης. Πάντως, όπως είπα, είμαι αρκετά ικανοποιημένο με το σχέδιο τη νομοδότηση και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με αυτά που προτείνει ο εισηγητή. Και ελπίζω να έχουμε ομαλή συνεργασία στη συνέχεια και να λάβω απάντηση στο ερώτημα τη παραφήνη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, είπε και ο εισηγητής της ΕΝΒΗ, είμαι σήμερα δύο σε ένα. Ε, ε, καταρχάς είμαι σκιώδης εισηγήτρια και έχω και παρατηρήσεις ε, του Νίλ Στόρβαλς, ο οποίος ευχαριστεί τον εισηγητή. Ναι, εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Άρχουτ για το σχέδιο γνωμοδότησής του. Ε, σε μεγάλο βαθμό η πρόταση αυτή διευκρινίζει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενισχύει τη διατύπωση σε κάποια σημεία. Το μοναδικό ε, μεγαλύτερο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ε, η η διαβριμένη ευθύνη του παραγωγού για τα αλλιευτικά εργαλεία. Ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει κάπως το θέμα αυτό. Άλλο θέμα είναι το κόστος ε, για τα συγκεντρωμένα απορρίμματα από τη θάλασσα. Ποιος θα πρέπει να καλύψει το κόστος αυτό. Δεν θέλουμε να ε, προσθέσουμε φόρτο στα αλλιευτικά σκάφη και τους αλλιείς. Ε, μπορεί λοιπόν νέα μέτρα να περιπλέξουν τα θέματα. Προσλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με τον εισηγητή ε, και με τους άλλους κοιώδεις εισηγητές στο ίδιο θέμα. Αυτά ήταν οι παρατηρήσεις του Νίλ. Τώρα θα σας παρουσιάσω τις δικές μου παρατηρήσεις. Όλοι φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται να ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να ομολογήσω ότι όλοι, όλοι οι παρόντες βρίσκουν, ε, ε, γνωρίζουν μάλλον ε, ότι είχα ασχοληθεί με τα πλαστικά στους ωκεανούς και ότι έμω το γνωρίζει αυτό. Είχαμε λοιπόν πολύ χρόνο να εξετάσουμε τα θέματα αυτά των ωκεανών και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν θα μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα με την οδηγία αυτή, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα θέματα, πρέπει να καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες. Αλλά στη συγκεκριμένη οδηγία, στην πρόταση αυτή, επικεντρωνόμαστε κυρίως στο τμήμα που αφορά την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Όπως ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να έχουμε σύστημα επιβράβευσης και όχι κυρώσεων όσον αφορά τη συλλογή απορριμμάτων από τη θάλασσα. Επίσης, ε, η απώλεια αλλιευτικών εργαλείων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι μπορεί να ε, δημιουργήσει πολλές ζημίες στο περιβάλλον, διότι συνεχίζεται η αλία χωρίς να γνωρίζει κανείς ε, τι ακριβώς ε, έχει αλλιευθεί. Εγώ θα ήθελα επίσης να μειώσω περισσότερο τα απόβλητα πάνω στα σκάφη, να έχουμε καλύτερο πλαίσιο για τα πράσινα σκάφη. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους ιδιοκτήτες πλοίων να μειώσουν τα απόβλητα. Επίσης, προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων με τους συναδέρφους μου στην Τραν ε, και εδώ, βέβαια, ναι, δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια εδώ πέρα, αλλά εντάξει, ο Νίλσε κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Γνωρίζω το θέμα της Μάρπολ και εδώ ακριβώ μπορεί να υπάρχει η δυσκολία, διότι η Μάρπολ είναι διεθνής και στόχος της είναι η περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν προστατεύει πάντα το περιβάλλον. Και γνωρίζουμε φυσικά ότι από πλευρά τη Ευρώπη δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα σε διεθνές επίπεδο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προχωράει κάπως παραπέρα. Ε, αναφέροντας, για παράδειγμα, τα υγρά απόβλητα, ε, θα πρέπει όμως το νερό από τη, τον καθαρισμό των δεξαμενών, αλλά πρέπει να εξετάσουμε γενικά τα υγρά απόβλητα. και γνωρίζω ότι άλλο η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άλλο η διεθνής νομοθεσία, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τη Μάρπολ. Πάντως σας ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή και είμαι βέβαιη ότι και από την Επιτροπή Τραν και από την Επιτροπή Ένβη θα ε, καταβληθούν προσπάθειες ώστε να προσπαθήσουμε να, πιέσουμε, να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει για πιο αποτελεσματική λύση σε διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω. Εάν έχουμε ε, μη ειδικά τέλη κατά 100% αυτό θα οδηγήσει σε συζήτηση, διότι από τη μία εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό να ακολουθήσουμε αυτή την οδό, από την άλλη δεν μπορώ να κρίνω τον όγκο των επικίνδυνων απόβλητων, ε, θα ε, αρνηθούν ε, παραλαβή οι λιμένες, ε, μήπως θα υπάρξουν αντιστάσεις. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι προβλήματα υπάρχουν. Πάντως γενικά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι πιο καθαρές θάλασσες και πιο καθαρούς λιμένες και αυτό επιθυμούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους κοιόδη εισηγητέ και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπονοφέ, ευχαριστώ. Με το πακέτο της κυκλικής ε, οικονομίας ε, που τώρα έχει γίνει νόμος, είδαμε πως ε, είναι σημαντική μια ορθή διαχείριση των αποβλήτων και για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη. Από τη σκοπιά αυτή δεν κάνουμε εξαίρεση για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία και έχουν και ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Στην περίπτωση των πλοίων έχουμε ζημίωση του περιβάλλοντος, αλλά και τις βιοπικιλότητας της πανίδας και της κλωρίδας. Είναι λοιπόν ε, ε, απαραίτητο θεμελιώδες οι λιμενικές εγκαταστάσεις να φέρουν τις κατάλληλες υποδομές. Επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε και πραγματικά πράσινα πλοία και να προλαμβάνουμε την παραγωγή αποβλήτων επί των σκαφών. Ένα άλλο σημείο είναι ότι δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε συστημικά αντικίνητρα το χάρη με ειδικά τέλη. Ειδικά τέλη που δεν μπορούν ε, να επιβαρύνουν τα λευτικά σκάφη, ε, τα οποία στα δίχτυα τους ε, πραγματικά συλλέγουν τα πάντα και ε, φυσικά πρέπει και να επερτρωθούμε περισσότερο στο να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Όμως θέλω να αναφέρω ένα πειραματικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Τοσκάνη και λέγεται Καθαρό Αρχιπέλογος ε, και θα παρουσιαστεί εδώ στο Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και από αυτό το πρόγραμμα ε, μέσα σε δύο μήνε έχουν συλλεχθεί 650 κιλά ε, σκουπιδιών στη θάλασσα από πέντε σκάφη. Και δύο είναι εναλλακτικέ ή θα τα φέρουν ε, ε, στα λιμάνια και θα πληρώσουν το τέλος τα σκάφη ή θα τα ξαναρίξουν στη θάλασσα. Λοιπόν, λοιπόν ευχαριστώ τον Σίτη που έχει αναφέρει αυτή την πτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την διαχείριση αυτών των αποβλήτων να την έχουν τα κράτη-μέλη και να προσπαθήσουμε να βρούμε και εναλλακτικέ ε, χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι με κανένα τρόπο οι αλληλεί ε, που συμμετέχουν ενεργά στην ε, παθητική αλία θα πρέπει να θεωρηθούν ω κάτοχοι των αποβλήτων και να του επιβάλλονται πρόστιμα γιατί κάτι τέτοιο δεν θα προωθούσε μία ενάρετη συμπεριφορά που κατά την άποψή μου θα πρέπει να υποστηριχθεί. Σας ευχαριστώ. Thank you. And now, uh, time Ευχαριστώ για την Κομισιόν. Η κυρία Κουτσόνσικα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Κατερχήν, σας ευχαριστώ για όλα τα θετικά σχόλια σε σχέση με την πρόταση. Επίσης ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΝΒΗ που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, γιατί πρόκειται για μια νομοθετική πρόταση που όντως αν και έχει νομική βάση στις μεταφορές έχει και μια πολύ ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση και περιβαλλοντικό στόχο να μειωθούν ε, τα απόβλητα και οι απορρίψεις των πλοίων στη θάλασσα και κυρίως ό,τι αφορά τις απορρίψεις σκουπιδιών. απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας, αλλά θα αναφερθώ και στην έκθεση του εισηγητή. Είναι καλό που ακούμε και σε αυτή την Επιτροπή, όπως και στην Επιτροπή Τραν, την ε, καθολική υποστήριξη στην αρχή αυτής της οδηγίας ε, με την προσέγγιση μη ειδικού τέλους. Γιατί πράγματι χρειαζόμαστε κίνητρα. Δεν αρκεί να πούμε ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτονται τα απόβλητα στάσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα καθιστά εύκολο και αποτελεσματικό. Ε, έτσι λοιπόν, εξού και η παροχή κινήτρων με την προσέγγιση του έμεσου τέλους, μη ειδικού τέλους, αλλά ταυτόχρονα καλούμε και για την ύπαρξη των κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. Φυσικά, ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι αρκετά απαιτητικό. Ε, φυσικά θα υπάρξει και το σύστημα ανάκτησης του κόστους ε, που θα βοηθήσει τους λιμένες να βελτιώσουν την ποιότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής που έχουν. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς έγιναν πολλές αναφορές εδώ, στην Σύμβαση Μάρπολ στο διεθνέ πλαίσιο. Ε, Μάρπολ ε, αφορά την ε, πρόληψη της απόρριψης αποβλήτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της παράδοσης των αποβλήτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Με την οδηγία αυτή δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως τι συμβαίνει στην ανοιχτή θάλασσα. Λεχθέντος αυτού, και ακούσαμε και από τον συγητή ότι αυτή η έννοια ε, έχει να κάνει και με την ε, ποινικοποίηση των ε, πλοίων που ρηπαίνουν σε ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει νομικό μέσο να το κάνουμε αυτό και καλωσορίζουμε τις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση για να τροποποιήσουμε και άλλα νομοθετήματα, δηλαδή να ποινικοποιήσουμε τα πλοία που ρηπαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Πολλές ερωτήσεις πάντοτε σε σχέση με τα λευτικά σκάφη. Καταρχήν, το να συμπεριλάβουμε τα λευτικά σκάφη στο έμεσο τέλος έχει ως στόχο να επιτρέψει στα λευτικά σκάφη να ενθαρρυνθούν να παραδίδουν χωρίς προς το κόστος ε, όλο αλλιεύουν στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό και συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει ώστε να πληρώνουν τελευταία σκάφη για όσα παραδίδουν. Ταυτόχρονα όμω, θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά αν αυτό είναι το κατάλληλο μέσο, το κατάλληλο εργαλείο για να εξετάσουμε όλα τα οικονομικά κίνητρα που θα αφορούν ε, μόνο τα λευτικά σκάφη, ε, παραδείγματος χάρη διάφορα προγράμματα ή τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλίες. Αυτή είναι το τομή, πιθανότητα που θα έπρεπε να εξετάσουμε περισσότερο, έτσι ώστε να δούμε ε, ότι αν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποια εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη για να καλύψουν το κόστος. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έχουμε στο παράρτημα 4 είναι τετρευπρόσδεκτο σε σχέση με τα έσοδα. Η έννοια του πράσινου πλοίου. Είναι σίγουρα κάτι που θα θέλαμε να αναπτύξουμε περισσότερο, όμως είναι μια έννοια που χρήζει της σας προσοχής. Γιατί θα πρέπει να ε, γίνει με, πλήρε, πλήρες τρόπο και θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλα είδη υποβλήτων όχι μόνο αυτά που έχουμε στο παραρτήμα 5. Γι' αυτό αρχικά προτείναμε να έχουμε εκτελεστική πράξη, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, γιατί ε, αν θα έχουμε την έννοια του πράσινου πλοίου, τότε να ε, λειτουργεί έτσι όπως πρέπει και να αφήσει τα πλοία να γίνουν πιο πράσινα. Υπήρχε μια ερώτηση ε, σε ό,τι αφορά ε, τα νερά αποστράγγισης, αυτά συμπεριλαμβάνονται. Επίσης ε, θα ελέγξουμε για την απάντηση στην ερώτηση ε, έρχεται σε σχέση με τις δεξαμενές. Ξέρω πάντα ότι το λέμε, αλλά τώρα είναι. Έρχεται. Θέλουμε να δούμε πόση επιρροή μπορούμε να έχουμε στις ε, αλλαγές στη σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ελπίζουμε θα γίνει τον Οκτώβριο είναι ότι θα υποβάλουμε εμείς κάποια στοιχεία σε σχέση με τα ε, θαλάσσια απόβλητα ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε φυσικά να αναφερθούμε και στο θέμα της παραφήνης. Όμως, ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μακρόχρονες, ε, όμως μπορούν να συμβούν αυτές οι τροποποιήσεις αν έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο ε, για να προστατεύουμε το διεθνές περιβάλλον, πρέπει να το, το θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να το κάνουμε μέσω διεθνών συμβάσεων. Γιατί μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει στα λιμάνια και μέσω του καθεστώτος επιβολής. Αλλά αν ε, δεν έχουμε ένα διεθνές ε, νομοθέτημα, τότε δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε ε, στο να έχουμε καθαρές θάλασσες και ωκεανούς στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Συγγνώμη, για τις πλατφόρμες που είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι πολύ πλοκό αυτό το θέμα γιατί στη Μάρπολ οι πλατφόρμες offshore, ανοιχτές θαλάσσης, θεωρούνται ως ορισμοί πλοίων. Όμως ε, θα ήταν συνεκτικό να συμπεριλάβουμε και τα πόβλητα από αυτές τις πλατφόρμες ε, στην οδηγία. Υπάρχουν όμως κάποια νομικά ζητήματα, κάποια νομικά ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και κατόπιν των συζητήσεων ελέγχουμε για το αν αυτά τα νομικά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν μπορούν να επιληθούν. Κάποιε από τι δυσκολίε είναι ότι όταν συλλεχθούν αυτά τα απόβλητα από μια πλατφόρμα, θεωρείται ότι δεν είναι απόβλητα που έχουν παραχθεί σε πλοίο, αλλά είναι απόβλητα υπομεταφορά. Transported waste, έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία. Σας ευχαριστούμε όμως για την ε, στήριξή σας και ανυπομονούμε να εργαστούμε με τις Επιτροπές ε, Περιβάλλοντος, Ελίας και Μεταφορών για να έχουμε μια καλή λύση σε σχέση με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο γρήγοροι. Ελπίζω ότι ο κύριος Εχάουτ δεν θέλει πάλι το λόγο. Κοιτάξτε, έχουν προβλεφθεί 45 λεπτά. Όχι, όχι, σύντομα θα είμαι. Πρώτα, πρώτα, πολλές ευχαριστίες όλους τους σκιώδες και την ε, για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, ε, δύο πραγματάκια για όσα αναφέρθηκαν. Πρώτα, πρώτα, για τις ε, πλατφόρμες. Θεωρούμε ότι πρέπει να καλύπτεται ε, και το φυσικό αέριο, είτε επιπλέει πλατφόρμα, είτε είναι σταθερή. Τέλος πάντων, ήδη τα είπαμε και θα συνηθούμε και περαιτέρω για να εξασφαλίσουμε το ότι είναι στεγανό νομικά το κείμενο και βγάζει νόημα και να τα καλύψουμε όλα. Τέλος πάντων θα το κοιτάξουμε και όπου χρειάζεται θα βελτιώσουμε την πρότασή μας. Όσον αφορά το πράσινο πλοίο θα το δούμε με την Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο το θέμα. Αποτελεί κίνητρο για πολλούς που δουλεύουν πάνω στα σκάφη να ξέρουν να διαχειριστούν τα απόβλητα. Μπορεί να είναι επίσης κίνητρο και για χαμηλότερο τέλος, άρα πρέπει να το θεσπίσουμε αυτό και να δούμε αν αρκεί ή όχι η εφαρμοστική πράξη επίσης ε, για το ηλεκτρονικό, την ηλεκτρονική αλληλεία τα είπαμε και ευχαριστούμε την κυρία Μποναφέ. If we are specifically with παθητική, συγγνώμη, πρόκειται για την παθητική αλία. Να δούμε μήπως τελικά δεν πρόκειται για κίνητρο εδώ ε, και τελικά να κανείς να εκφορτώνει αυτά τα οποία έχει ελεύσει κατά το αυτό το τρόπο τη παθητική Και προβληματίζεται και η Επιτροπή να δούμε και με την εισηγήτρια ποιες θα είναι οι εθνικές αρμοδιότητες να το δούμε για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο με, με τέλη το σκάφος. Ωραία, ωραία είναι που συμφωνείτε για τις τροπολογίες όταν αυτή την ποινικοποίηση για το PPR. Μας τα είπατε ως σκιώδης ηγήτρια, είναι αλήθεια ότι αυτά τα γράψαμε πριν διαμορφωθεί η πρόταση για την ε, ενιαία μοναδική χρήση. Ε, γι' αυτό το, το γράψαμε. Τώρα περιέχεται εκεί. Δεν πειράζει. Αφού είναι αλλού, ας το βγάλουμε. Το θέμα είναι κάπου να υπάρχει μία ρύθμιση. Πλαστικά μια χρήση αφού καλύπτεται από εκεί, εντάξει. Γι' αυτό το βάλαμε. Ποιο ξέρει, μπορεί και να συμβάλαμε έτσι να το βάλει η Κομισιόν στην πρότασή τη. Σα τα πάω όσο πιο σύντομα μπορούσα, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Βλέπετε, έχουμε τώρα χρόνο να δούμε το δεύτερο ημίχρονο τον αγώνα παίζεται τώρα. Όχι, όχι, δεν παίζει η Ολλανδία. Και σας ευχαριστούμε. Έχουμε 28 Ιουνίου ως προθεσμή για τις τροπολογίες και 14 Σεπτεμβρίου θα γίνει η ψήφιση στην Τραν. 9 Οκτωβρίου και ελπίζουμε στην ε, Ολομέλεια τη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Νομίζω, ελπίζω τελειώσαμε. Καλή ξεκούραση.